Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα το απόγευμα με τη συνάντηση της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον, τον Αντιπρόεδρο κ. Ντομπρόσκη στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου. Είναι η δεύτερη φορά που τα λέμε φέτος και να σας υπενθυμίσω πως τα ζητήματα για σήμερα είναι η οικονομική σταθερότητα και η ένωση κεφαλαίου αγορών, όπως επίσης και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα, οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ και θα το υπενθυμίσω ευγενικά να περιοριστείτε σε αυτά τα θέματα κατά τι ερωτήσει. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Αντιπρόεδρο για να ξεκινήσει με κάποια εισαγωγικά σχόλια και μετά να σας υπενθυμίσω αγαπητοί συνάδελφοι πως σήμερα πέντε λεπτά ο καθένας. Οπότε ρωτάτε, σας απαντούν και αν έχετε χρόνο μπορείτε να επανέλθετε. Όμως σας παρακαλώ πολύ ε, να ε, σηκώνετε το χέρι σας έτσι ώστε να το ξέρω για να σας ξαναδώσω το λόγο. Λοιπόν, χωρίς να καθυστερώ, ο λόγος την Πρόεδρο. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στη δική σας επιτροπή, έτσι ώστε να μιλήσω για την δουλειά που κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να είναι πιο δυναμική, πιο ολοκληρωμένη και πιο ισόρροπη η χρηματοπιστωτική αγορά στην Ευρώπη. Από την τελευταία φορά που τα είπαμε έχουμε προχωρήσει έτσι ώστε η, η, Ένωση Κεφαλαιογορών μέχρι το 2019 να έχει κλείσει, να κλείσουμε και το θέμα της Τραπεζικής Ένωσης και να δημιουργήσουμε ένα πιο αθεκτικό πλαίσιο για το χρηματοπιστωτικό κλάδο. Εμείς Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε και στο εσωτερικό και με τους διεθνείς εταίρους έτσι ώστε να έχουμε ίσους κανόνες παιχνιδιού για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Ποιες είναι οι προκλήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό. Καταρχήν, διαπραγματεύσει το Brexit ξεκίνησαν χτες. Οπότε φτάνει η ημέρα όπου το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό κέντρο της Ευρώπης θα αποκοπεί από τους 27. Και παρόλο που αναπτύσσεται η οικονομία, αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια προβλήματα που δεν μας επιτρέπουν να ανακάμψουμε όσο θέλουμε. Δηλαδή, υψηλά επίπεδα χρέου, χαμηλή παραγωγικότητα και μια συνεχής έλλειψη μακροπρόθεσμη επένδυση στι επιχειρήσει και στι πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών. Χωρί το ε, Ηνωμένο Βασίλειο, η αγορά μετοχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και πάλι το 15% τη κεφαλοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά η κατάτμιση δεν επιτρέπει στο χρηματοπιστωτικό μα κλάδο ε, ε, να αποδείξει πόσο δυναμικό είναι. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα στεναρότερο, ασφαλέστερο και πιο καινοτόμο χρηματοπιστωτικό κλάδο μέσω τη ολοκλήρωση. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν οι δικέ μα χρηματοπιστωτικέ αγορέ να αναπτυχθούν σε όλη την Ευρώπη, να είναι πιο παραγωγικέ και να δημιουργήσουν θέσει εργασία. Επίση, διασυνοριακέ χρηματοπιστωτικέ ροέ στην χώρο του ευρώ είναι κομβικό σημείο για να έχουμε καλύτερη μετάδοση των νομισματικών μα πολιτικών και για να μπορέσουμε να αποβροφήσουμε τα μη συμμετρικά σοκ. Επίση, μεγαλύτερη ε, καινοτομία μια περισσότερη κοινοτομία και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα big data και τις δυνατότητες της fintech ε, είτε σε μικρές είτε σε μεγάλες αγορές είτε σε μερίδια αυτών. Να σας πω πως αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε το χρηματοδοτικό μας ε, κλάδο ε, για να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Και αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μεγάλα εμβληματικά project και θέλουμε να μας στηρίξετε εσείς για να περάσουμε από εκεί που είμαστε σήμερα σε εκεί που θέλουμε να βρεθούμε στο μέλλον. Να ξεκινήσω λοιπόν να μιλήσω ε, μιλώντας για την Ένωση των και αγορών κεφαλαίων. Καταρχήν, με τη δική σα βοήθεια, για να έχουμε μια τέτοια ενιαία αγορά, μας στηρίξατε εσείς, έχουμε κάνει πρόοδο με το σχέδιο δράση και ε, πετύχαμε μια συμφωνία επί τη αρχή για ε, τιτλοποίηση, η οποία θα είναι ασφαλή και διάφανη μαζί σα, Να συγχαρώ τον Πολ και τον του Μορκάρας, για την συμφωνία αυτή που μπορεί να ξεκλειδώσει γύρω στα 150 δι σε δανειοδοτήσει για νοικοκυριά και εταιρείε. Επίση θα ήθελα να ευχαριστήσω την σύρπα ποιετικά είναι για τη δουλειά που έχει κάνει, έτσι ώστε να έχουμε πολιτική συμφωνία για τους κανόνες, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα χρήματα και για τα επενδυτικά κεφάλαια κινδύνου και για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και έχουμε τώρα μέχρι 400 ε, εκατομμύρια ευρώ που θα τα κινητοποιήσουμε έτσι ώστε να μοχλεύσουν πάνω ε, γύρω στο 1,6 δις ε, πολύ σύντομα. Και θα ήθελα να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γρήγορα να κλείσει τι τυπικέ διαδικασίε, έτσι ώστε να δρέψουν τα πλεονεκτήματα όλων αυτών οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έχουμε την, ε, το σχέδιό μας λοιπόν για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Αυτή τη στιγμή είναι στο μεσοπρόθεσμο σημείο και έχουμε κάνει ε, τα δύο τρίτα της διαδρομής σε σχέση με το σχέδιο δράσης του 2015. Πρέπει όμως να χρησιμοποιήσουμε τις επιτυχίες μας και να προχωρήσουμε ώστε να έχουμε περισσότερη ολοκλήρωση ενώ του 2019. Θέλω να με στηρίξετε παραπάνω και πρέπει να σας πω ότι στην αναθεώρηση αυτής της Ένωσης έχουμε προτείνει κάποιους στόχους. Για παράδειγμα, να διευκολύνουμε τις μικρομεσαίες που ζητούν κονδύλια στις ε, δημόσιες αγορές, πώς ελαφρύνοντας τις κανονιστικές διατάξεις που βαρύνουν. Θέλουμε να έχουμε συνεκτική εποπτεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη δημόσια διαβούλευση για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές λάβαμε πάνω από 220 απαντήσεις από μία σειρά ενδιαφερομένων και θα ε, δρομολογήσουμε τις εξελίξεις σύμφωνα με τα ευρήματα του φθινόπωρα. Αυτή τη στιγμή για την αδειοδότηση και για τα διαβατήρια, για τις δραστηριότητες χρηματοπιστωτικής τεχνικής, fintech δηλαδή, ε, ζητάμε το ποιο θα είναι το πλαίσιο. Θέλουμε οι καινοτόμε εταιρείε να δημιουργήσουν μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, να μείνουν στην Ευρώπη και να είναι παγκόσμια ανταγωνιστικέ. Και επίση θέλουμε να δούμε τι γίνεται με την αγορά των πράσινων ομολόγων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομάδα υψηλού επίπεδου που προετοιμάζει κάποιου είδους ε, συμβουλές έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα να τις εντάξουμε στους χρηματοπιστωτικούς κανονισμούς και να συνεχίσουμε από εκεί το πρώτο τρίμηνο του 2018. Επίσης, για το νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή μιλάμε ε, για τα καλυπτόμενα ομόλογα για, μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και όπως και επίσης για τις ιδιωτικές συντάξεις που θα λειτουργήσουν ως ε, προϊόν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά για το προηγούμενο και το επόμενο είναι η ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Να σας πω πως έχουμε πάρει μια σειρά από προτάσεις και θα τις βάλουμε ε, στα σκαριά έτσι ώστε να λύσουμε και τα προβλήματα της αγοράς παραγόγων. Γιατί ξέρετε πως εκεί βρίσκουμε εκατομμύρια τρισεκατομμυρίων ε, ευρώ. Είχαμε μια πρόταση τον Νοέμβριο για τους κεντρικούς αντισυμβαλώνους και ε, παρουσιάστηκε η πρόταση αυτή έτσι ώστε οι αρχές να έχουν ε, τα εργαλεία που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν την, ε, το μάλλον ε, άγνωστο σενάριο μιας χρεοκοπίας σε επίπεδο κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε και το πλαίσιο που θα αναθεωρήσει τις απαιτήσεις για τα παράγωγα, τα εξοχρηματιστριακά έτσι ώστε να δώσουμε πλεονεκτήματα και σε κάποιους αντισυμβαλόμενους που δεν είναι χρηματοπιστωτικές εταιρείες. Επίσης, τεχνικές λύσεις ε, μέσα σε τρία χρόνια έτσι ώστε οι μελλοντικοί συνταξιούχοι να δουν ότι προστατεύονται οι ε, Συντάξεις στο μέλλον. Επίσης, θέλουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στο θέμα αυτό των κεντρικών αντισυμβολωμένων και να δούμε πώς εμείς μπορούμε να προλάβουμε τις εξελίξεις. Καταλαβαίνετε πως για όλα αυτά το Brexit αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση και εμάς η πρότασή μας είναι να έχουμε μια πιο πανευρωπαϊκή εποπτική προσέγγιση έτσι ώστε τους κεντρικούς αντισυμβολόμενους να τους παρακολουθούμε ευρωπαϊκά με ένα διτό σύστημα έτσι ώστε να λαμβάνουμε υπόψη τι γίνεται και από τα μη ευρωπαϊκά, τα, τα κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράδειγμα αυτό που κάνουν οι ΙΠΑ σε επίπεδο εποπτείας και να σα πω πω ω τελευταίο καταφύγιο όταν χρειάζεται να εξασφαλίσουμε τη χρηματοσυντητική σταθερότητα οι αρχέ μπορεί να απαιτούν από μεμονωμένους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους ε, να εγκατασταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν θεωρούμε πω συστημικά είναι σημαντική. Και ελπίζουμε ότι και στου φακέλου αυτού θα μα στηρίξετε. Να περάσω τώρα στην, ε, στον τραπεζικό κλάδο. Καταρχήν χαιρετίζω το γεγονό πω ο Γκούνερ Χόκμαρ και ο Πίτερ Σίμων αυτή τη στιγμή εργάζονται πάνω στο πακέτο για τα τραπεζικά έτσι ώστε να είναι πιο ανθεκτικέ οι ευρωπαϊκέ τράπεζε. Την περασμένη εβδομάδα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν δύο σημαντικά κομμάτια του πακέτου. Κατα στην ιεραρχία των πιστωτών, το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούν οι μεγαλύτερες ε, τράπεζες θα μπορούν να παρουσιάζουν κάποια ε, στεναρά, ε, κάποιες στεναρές αντιστάσεις σε περίπτωση που έχουμε ε, bail-in, δημιουργώντας ε, κάποια κοινά ευρωπαϊκά στοιχεία ενεργητικού. Αυτό θα δώσει μεγαλύτερη σαφήνεια και θα τους βοηθά να κάνουν αξιολόγηση και τιμολόγηση κινδύνου. Επίσης, ΔΕΛΤΑ 9 Εδώ θέλουμε να δούμε τι γίνεται με τις μεγάλες εκθέσεις και θα ήθελα να παρακαλέσω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει γρήγορα έτσι ώστε τα κομμάτια αυτά του πακέτου να έχουν μπει στα, ε, και αυτά σε κάποια διαδικασία έγκριση μέχρι τα τέλη τη χρονιά. Επίση, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κλείσουμε και τι μεταρρυθμίσει τη Βασιλεία. Το να παρατείνουμε την αβεβαιότητα δεν είναι καθόλου καλό για το χρηματοπιστωτικό κλάδο. Οπότε οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει ε, να έρθει γρήγορα και μέσα σε αυτή την συμφωνία θα πρέπει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι στο θέμα του κινδύνου και να λάβουμε υπόψη κάποια ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα πώς χρηματοδοτείται η κατοικία, η στέγη ε, μέσω ε, ενυπόθηκων δανείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε τον κλάδο τον τραπεζικό έτσι ώστε να μην έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις απαιτήσει. Ε, ε, κεφαλαίων για τις τράπεζες. Επίσης, στο θεματολόγιο μας είπαμε ε, στεναρός ε, κλάδος, έτσι ώστε να έχουμε ένα πανευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, να δούμε τι γίνεται και με τα δάνεια των τραπεζών και να σας πω πώς από την κρίση και μετά κάναμε πολλά. Και η πρόσφατη λύση των προβλημάτων της Banco Popular στην Ισπανία έδωσε τίτλους εφημερίδες και κάναμε τη διαδικασία μέσω της Τραπεζικής Ένωσης, που είναι πλέον πλήρω λειτουργική, αλλά θα πρέπει μόλι καταλαγιάσει ο θόρυβο, να δούμε ακριβώ τι μπορούμε να ε, βελτιώσουμε. Επίση, υπάρχουν κάποια κομμάτια τη Τραπεζικής Ένωση που λείπουν. Πρέπει να τα στήσουμε έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη κατανομή του κινδύνου και στο μέλλον. Έχουμε μια ισόρροπη και σταδιακή πρόταση έτσι ώστε να έχουμε και ένα σύστημα ευρωπαϊκό ασφάλισης καταθέσεων και θα πρέπει να κάνουμε πρόοδο έτσι ώστε και αυτό να μπει στην Τραπεζική Ένωση. Και επειδή έχουμε και τον ενιαίο μηχανισμό επίλυση ε, κρίσεων που πρέπει να είναι πιο αξιόπιστο Σύπαμε είπαμε πως χρειαζόμαστε και εδώ ε, κοινού κανόνε που θα είναι αρκετά ε, ε, ευρύ έτσι ώστε να, να καλύπτουν πάρα πολλά σενάρια. Και κλείνω λέγοντα πώ θέλουμε να παγιώσουμε τη θέση μας ενώπιον στι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με τη δουλειά μα και θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ολοκλήρωση και να κλείσουμε με τα θέματα τη Τραπεζικής Ένωση και τη Ένωση Κεφαλαιογορών Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ για τι παρατηρήσει για τι τοποθετήσει σα και θα ακούσουμε του ομιλητέ ομιλητέ εκ μέρου των ομάδων. Τον κύριο Ματουσέλο πρώτα, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Έχετε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Μια ερώτηση. Και πληροφορίες θα ζητήσω μετά. Σχέση με ένα, μια επιστολή που σας έστειλαν πολλοί συνάδελφοι συνυπογράφοντας. Το ερώτημα λοιπόν. Έχουμε δει ότι στα προβλήματα των τραπεζών ενεπλάξαν οι ίδιοι οι πελάτε. Τα δεδομένα μα λένε ότι από το 2013 στο 2017 το κόστο των τρεχόντων λογαριασμών αυξήθηκε κατά περισσότερο από 17%, 115 ευρώ περίπου σε 135 ε, κατά μέσο όρο. Έτσι λοιπόν μπορεί να μην έγινε το Μπέιλιν ακριβώς, αλλά τελικά ο καταθέτης ο μικροκαταθέτης ε, πλήρωσε το κόστος ε, της ε, απρόσεκτης διαχείρισης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το κόστος αυτό λοιπόν το πληρώνει ο καταναλωτής που αποταμιεύει ο καταθέτης και βεβαίως αυξάνει το κόστος διαρκώς της διαχείρισης των τερχών των λογαριασμών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτού ορισμένες τράπεζες ζητούν την συμβολή αυτή, την οικονομική, στον καταθέτη, επιβάλλοντας μάλιστα ένα τέλος με τον τίτλο «Τέλος Μπέιλιν». Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν τέτοιο όρο, είναι σωστό αυτό. Και μάλιστα σας στείλαμε μια επιστολή για να περάσω στο επόμενο θέμα με υπογραφές πάνω από 40 συναδέλφων. Και ζητούσαμε της ε, θέσης σε σχέση με την καταναλωτική πίστη. Ένα προϊόν πολύ διαδεδομένο στην Ιταλία, με πολύ χαμηλό επίπεδο κινδύνου, όπου παρά το χαμηλό επίπεδο κινδύνου έχουν βάρο κινδύνου τα χρηματοπιστωτικά που χορηγούν, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χορηγούν αυτή την ε, καταναλωτική πίστη στο 85%. Υπάρχει τρόπος να κατέβει στο 35% ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να αποδεσμεύσουν κεφάλαια. Κεφάλαια τα οποία μετά μπορούν να διατεθούν ε, σε δάνεια στεγαστικής πίστης και γενικώ να βοηθήσουν ε, να αναπτυχθεί η οικονομία. Ο κύριος Δομπρόφσκης. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. περισσότερες από μία ερωτήση στην πραγματικότητα για το κόστος των τριχών λογαριασμών καταρχάς. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες, ε, θα σας πω, που οδηγούν στην αύξηση του κόστους των τρεχών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένου και του χαμηλού επιτοκίου, που εκδηλώνεται στο παρόν περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι τράπεζες. και αυτό προσπαθούν να ενισχύσουν αυξάνοντας τα διάφορα τέλη για τον καταναλώτη. Και αυτό το βλέπουμε και στους τρέχοντες λογαριασμούς. Στο βαθμό αυτό λοιπόν εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την υπηρεσία που προσφέρεται στον καταναλωτή μέσω του προγράμματος δράσης για τις λιανικές οικονομικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και διασυνοριακά με την παροχή προϊόντων στη διάθεση του καταναλωτή, βέβαια με καλύτερη ενημέρωση και δυνατότητα σύγκριση για τον τρόπο με τον οποίο ε, τιμολογούν τα διάφορα τέλη οι τράπεζες. και έτσι θα μπορεί ο καταναλωτής, ο καταθέτης έχοντας υπόψη το κόστος αυτό, τις εισφορές που του επιβάλλονται, να διαλέξει το προϊόν που προτιμά. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο έχει φτάσει τώρα στις νομικές μας υπηρεσίες για να ε, ολοκληρωθεί το σχέδιο δράσης. Για την αυτοδιάσωση, Μπέιλιν. Είναι κάτι το οποίο έχει επίσης συμφωνηθεί προκειμένου να προστατευθεί το συμφέρον του φορολογουμένου, ώστε να μην είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει πρώτος τις συνέπειες των σφαλμάτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. με υπερβολικό μπόνους και με κλιματικές ακόμη δραστηριότητες και θα πρέπει και οι επαγγελματίες επενδυτές, τους ενθαρρύνουμε τουλάχιστον, να ε, μεριμνούν ώστε να παρακολουθούν με προσοχή την διαδικασία και τις λειτουργίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο πνεύμα μιας χρηστής παγκόσμια χρηματοπιστωτική διαχείριση. Τώρα, για το δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με τις ε, με την καταναλωτική πίστη. Έχουμε λάβει την επιστολή σας όντως, την αξιολογούμε αυτή τη στιγμή. Βεβαίω πρέπει να ε, σημειώσω ότι η οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια του Κοινοβουλίου, άρα έχετε την ε, πρωτοβουλία. Πάντως αξιολογούμε την επιστολή σας και κατ' ουσίαν πρόκειται για ζήτημα αξιολόγηση των δεδομένων και τη στάθμιση του κινδύνου ανάλογα με το κάθε προϊόν. Θα κοιτάξουμε λοιπόν εάν τα δεδομένα που έχουμε στη θέσή μας επιβεβαιώνουν τον ε, ισχυρισμό ότι είναι χαμηλότερο το επίπεδο κινδύνου για αυτά τα προϊόντα σχέση με κάποια άλλα και θα σα απαντήσουμε. Ευχαριστώ κυρία Γκίλ, σοσιαλιστέ Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Θέλω να θέσω δύο θέματα. Πρώτον, στην παρουσίασή σας περιγράψατε τη μεταρρύθμιση της εποπτείας για να γίνουν πιο εύρωστοι η κεντρική αντισυμβαλόμενη, κάτι που θα ωφελήσει ευρύτερα καταναλωτές και επιχειρήσεις. Χαιρετίζω την ρεαλιστική σας στάση που τηρήσατε στην συνέντευξη τύπου πέρσι. Νομίζω ότι πράγματι υπάρχει ε, πλέον μια ε, πιο στενή συνεργασία μεταξύ των τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο, ε, μένει ανοιχτό το ζήτημα της μετεγκατάστασης των κεντρικών αντισυμβαλωμένων από το Λονδίνο στην Ευρωζώνη. Δεδομένου λοιπόν των στοιχείων που έχουμε στα χέρια μας, η, αντι... η των κεντρικών αντισυμβαλωμένων θα δημιουργήσει κόστος και θα πρέπει οι τράπεζες που θα επιλέξουν αυτή την επιλογή, θα επιλέξουν αυτή την, αυτό το δρόμο να ε, ανταποκριθούν σε υψηλότερα κριτήρια κεφαλαϊκής επάρκειας. Πρώτον. Δεύτερον, για να ολοκληρωθεί ε, αυτό ο φάκελος χρειάζεται να λειτουργήσει τόσο έντιμος διαμεσολαβητής διαπραγματευτής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οικονομική σταθερότητα και όχι μόνο να ε, εξασφαλιστεί το οικονομικό όφελος του ενός κράτους μέλους έναντι του άλλου. Επίσης, Κάνατε μια άλλη ανακοίνωση για, την βιώσιμη, για, τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και χαιρετίζω και το γεγονό ότι είπατε ότι πρέπει να επιτεθούν οι στόχοι για το κλίμα των Παρισίων. Ε, πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε ότι θα κατευθυνθούν δάνεια προς την πράσινη οικονομία με μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την κεφαλική επάρκεια και ότι θα ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στην πράσινη οικονομία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα ανταποκριθείτε σε αυτά τα καθήκοντα. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα λοιπόν. Ένα που αφορά την πρόσφατη πρότασή μας για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους από τρίτες χώρες και το άλλο για την βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πρώτον, πιστεύω ότι έχουμε ε, εξειδικεύσει την πρότασή μας και εξασφαλίζει πλέον τη χρηματοπιστική σταθερότητα ελαχιστοποιώντας ε, τις ζημίες για τις επιχειρήσεις. Προφανώς υπάρχει αντίκτυπος, κάναμε και μια μελέτη αντικτύπου που το καταδεικνύει αυτό, αλλά ο δρόμος που χαράξαμε ορίζει ότι οι αρχές μπορούν να λαμβάνουν μέτρα σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την χρηματοπιστική σταθερότητα απλά και μόνο με αυτά τα μέσα ε, τραπεζικής εποπτείας. Οι γνώμες λοιπόν σε αυτό το θέμα διήστανται. Και βλέπω ότι και εδώ στην Επιτροπή σας υπάρχουν Υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα απόψεων, να το πω έτσι. Ακούσαμε από τον Μάρκους Φέρμπερ ότι η Κομισιόν έχει χάσει το θάρρος της και ότι δεν χρειαζόμαστε κατά περίπτωση ανάλυση, αλλά έναν βασικό κανόνα ότι η καθάριση θα πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. ακούσαμε και άλλη άποψη, την αντίθετη. Ότι η ανάλυση στο ευρωπαϊκό πλήσιο θα, όπως είπε η κυρία Σουίνμπορν, θα αντίκειτο στην, ε, στον στόχο το, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της εξασφάλισης της. Σταθμίσαμε πολύ προσεκτικά όλες τις απόψεις. Όσον αφορά τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και το ρόλο που μπορεί να παίξει ε, ο ιδιωτικός τομέας στην επιτεύξη των στόχων του Παρισιού. Στην ενδιάμεση αναθεώρηση της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών, ε, στο πλαίσιο αυτής της ενδιάμεσης αναθεώρησης, περιμένουμε να εκδοθεί ε, μια σχετική μελέτη και μάλιστα τον Ιούλιο θα γίνει και μια ευρύτατη διαβούλευση εδώ στις ε, Βρυξέλλες, ενώ η οριστική ενδιάμεση έκθεση αναμένεται να εκδοθεί το Σεπτέμβριο. Αν, δείτε όμως τα ποσά ε, που χρειάζεται να επενδυθούν για να επιτεθούν οι στόχοι του Παρισίου για τους δύο, δύο βαθμούς Κελσίου, βλέπετε ότι αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με δημόσια χρήματα, χρειάζεται και, χρειάζονται και ιδιωτικά κεφάλαια και αυτόν τον στόχο υπηρετεί η, η δική μας δράση. Ευχαριστώ. Ε, εκ μέρους του ECR θα σας θέσω εγώ ε, ερωτήματα. Προφανώς και εγώ θα αναφερθώ στα, στο ζήτημα των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Από την ε, περίοδο του ξεσπάσματος της ε, οικονομικής κρίσης, οι G20 είχαν πει ότι αυτό το θέμα θα αποτελέσει βασικό κλειδί για την επίλυση ε, των προβλημάτων που ε, παρουσιάστηκαν στην, στην, για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Και πράγματι φαίνεται ότι το βρετανικό μοντέλο ε, γίνεται παράδειγμα προς μίμηση. Γι' αυτό και με ανησύχησε κάπως η πρότασή σας. Μπορείτε να, μας διασφαλίσετε ότι η κεντρική εκαθάριση ε, και η αμοιβαιοποίηση του χρέους εξακολουθεί να είναι ο, ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να επιλύουμε τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Και ε, Ποιο ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών κατά την εκτέλεση των εποπτικών τους καθηκόντων. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν μια εθνική αρχή και η ΕΣΜΑ αποφασίσουν ότι ένας Ευρωπαίος κεντρικός ε, πρέπει να ε, συμμορφωθεί με μια απόφαση, ε, τότε κάθε κεντρική τράπεζα της Ευρώπης μπορεί να ασκήσει βέτο σε αυτή την, ε, σε αυτή την απόφαση. Για παράδειγμα, για το, το, το ουγγρικό χρέος ε, ε, μπορεί σε αυτή την περίπτωση, αν, αν αυτό τεθεί ως θέμα, μπορεί η Ουγγρική Κεντρική Τράπεζα να ασκήσει βέτο με αποτέλεσμα να θέσει κίνδυνο για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αυτή είναι και η δική σας ερμηνεία ε, όσον αφορά τα ζητήματα της χρηματοπιστικής σταθερότητας γιατί θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε, διαφορετικοί τρόποι χειρισμού των θεμάτων της χρηματοπιστικής σταθερότητας από τις κεντρικές τράπεζες. Για το ερώτημα αυτό, πρώτον να σας διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν εξακολουθεί να επιδιώκει αποτελεσματική λειτουργία των παγκόσμιων περιστατικών αγορών. Και όταν οι παγκόσμιοι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι ενδέχεται να θέσουν να απειλήσουν την ε, ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Η πρόταση της Κομισιόν με άλλα λόγια μας επιτρέπει να εξετάσουμε τους κινδύνους αυτούς και να ανταποκρινόμαστε ανάλογα. Ε, και στόχος μας είναι να θεσπίσουμε όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες ώστε και οι εκδότες τράπεζες να έχουν ε, λόγο στη διαχείριση αυτών των ε, υποθέσεων. Συγγνώμη, να επανέλθω. Συγκεκριμένα. Όσον αφορά τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών φαίνεται σαν να έχουν ηγετικό ρόλο. Θα πρέπει οι κεντρικές τράπεζες λοιπόν να τίθενται επικεφαλής της διαχείρισης προβλημάτων στη χρηματοπιστική στάθερα. Ο ΕΣΜΑ και η, και η Κεντρική Τράπεζα τίθενται επικεφαλής προκειμένου να εξορροπούνται οι διαφορετικές απόψεις ή προσεγγίσεις. Κάποιες φορές μπορεί να απαιτείται η εξέβρεση κάποιου, κάποιας ισορροπίας. κύριος Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Ντομπρόσκης, αγαπητοί συνάδελφοι. το χρέος, το κυβερνητικό, δεν είναι ακίνδυνο και δεν θα πρέπει να το μεταχειριζόμαστε ως κάτι ακίνδυνο στους δικούς μας κανονισμούς. Και ξέρετε, όπως το ξέρει και το Δουνουτού και το Εποπτικό Συμβουλίο και η ΕΚΤ, ε, πως ισχύει αυτό που λέω. Εσείς το δέχεστε και ποια μέτρα θα λάβετε. Θα καταθέσετε νομιθετική πρόταση για το θέμα του ε, κρατικού χρέους το οποίο είναι μη ασφαλές στοιχείων ή όχι. Και επίσης, συγκέντρωση του χρέους, ε, του κεντρικού χρέους, του κρατικού χρέους σε λίγα χέρια. Διπλασιάστηκε το ποσοστό στην Ισπανία, πολλαπλασιάστηκε στην Ιταλία. Ανισορροπία μεταξύ ε, ιδιωτικών τραπεζών και κρατικών τραπεζών. Πολύ επικίνδυνα όλα αυτά σε στιγμή θα το αντιμετωπίσετε? Θα έχουμε όρια ανοίγματο στο κρατικό χρέος για τους ιδιώτες δανειστές ή όχι. Okay. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε το θέμα ε, μιλάμε για την εμβάθυνση της ε, ΟΝΕ και εκεί κάνουμε όλες αυτές τις σκέψεις, αλλά γίνονται σε δύο φάσεις τα όσα προβλέπονται. Καταρχήν έχουμε την πιο άμεση φάση, όπου είμαστε πιο περιγραφικοί και πιο συγκεκριμένοι για το τι πρέπει να γίνει και μια δεύτερη φάση που είμαστε πιο ανοιχτοί και παρουσιάζουμε κάποια αναλλακτικά σενάρια τα οποία θα μπορούσαν να επιλέξουν τα κράτη-μέλη και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Οπότε, βράχη πρόθεσμα προτείνουμε να βασιστούμε στα όσα έχει κάνει ε, το Συμβούλιο για το Συστημικό Έλεγχο, ε, έτσι ώστε να έχουμε καλύψει όλα τα θέματα αυτά με τα κρατικά ομόλογα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ούτε αμοιβαιοποίηση, ούτε σύνδεση κρατικών ομολόγων με συγκεκριμένες κατηγορίες επικινδυνότητας. Άρα λοιπόν αυτό δεν θα το βρείτε στην πρότασή μας. Για τη δεύτερη φάση που ακόμα βρίσκεται πιο πολύ σε επίπεδο σκέψης, αναρωτιόμαστε τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να θεωρηθεί ε, ασφαλή, ε, τι, μπορεί να είναι ασφαλή στοιχεία ενεργειακού, ε, ενεργητικού στην Ευρώπη, τι γίνεται με την τιτλοποίηση και ποιο θα πρέπει να είναι η κανονιστική αντιμετώπιση του κρατικού χρέους. Το θέμα πάντως βρίσκεται στο τραπέζι. Τώρα, για τα ανοίγματα σε κρατικό χρέος, όντως, αυτό είναι ένας τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε, δηλαδή για την περίπτωση που έχουμε αυτές τις υπερβολικές εκθέσεις, αλλά αυτό που προτείνουμε δεν είναι περιθω, ε, ε, περιορισμοί, ε, κατόφλια ή οροφές στο άνοιγμα, αλλά ο κρατικά ομόλογα τα οποία καλύπτονται από εγγυήσεις, το οποίο σημαίνει ότι μπορούν αυτές οι εγγυήσεις να τις αποκτήσουν οι τράπεζες. Πώς? Με έναν τρόπο που αμέσως διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό τους, έτσι ώστε να έχουν μικρότερο άνοιγμα στα δικά τους κρατικά ομόλογα. Δηλαδή είναι ένα προϊόν που απευθύνεται στις ευρωπαϊκές τράπεζες, μπορούν να το αποκτήσουν, που επιτρέπει τη διαφοροποίηση μέσω αυτών των εγγύησεων. 30 ερωτήσεις, 30 δευτερόλεπτα με συγχωρείτε, έχω όχι 30 ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας, αλλά πείτε μου εσείς τι πιστεύετε για το θέμα που έθεσα. Είναι ακίνδυνο το κρατικό χρέος ως στοιχείο ενεργητικού ή όχι. Δεν θέλω να δημιουργήσω σύγχυση. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Δεν θέλω εγώ να αυτοσχεδιάσω τώρα εδώ. Ξέρετε ποια είναι η τρέχουσα μεταχείριση. Συνδέει μηδενικούς συντελεστές επικινδυνότητας. Όταν προχωρήσουμε λοιπόν σε μη μηδενικούς ε, συντελεστές ε, επικινδυνότητας για το κρατικό χρέος, το οποίο το έχουμε ε, ως εναλλακτική, τότε, στο έγγραφό μας, τότε θα πρέπει να έχουμε και τα απαραίτητα χέγγια και εγγυήσει έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα σε χώρες οι οποίες ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν αυτό το σενάριο. Θα ήταν πιο εύκολο λοιπόν να ξεκινούσαμε όλοι από μηδενική βάση. Δυστυχώς όμως αυτό δεν συμβαίνει. Ξεκινάμε από εκεί που είμαστε όλοι σήμερα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι σημαίνει η χρηματοπιστική σταθερότητα και ποιες είναι οι συνέπειες αυτής. Αυτό ακριβώς έχουμε τοποθετήσει στο έγγραφο. Κύριε Τρεμόσα, θεωρείτε πως ήταν απάντηση μονολεκτική. Πέντε λεπτά λοιπόν τα κλείσατε. Κύριε Παπαδημούλη, γκουε. Oh, you did perfect. Uh, Mr. I will speak in Greek, so please use your headphones. Θα μιλήσω ελληνικά, οπότε παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στην Επιτροπή μας, κύριε Αντιπρόεδρε. Σημείωσα με ενδιαφέρον ότι επισημάνατε την ανάγκη να ολοκληρωθεί η, η τραπεζική ενοποίηση και η Ένωση των Κεφάλαιων Αγορών αλλά έχει και ένα τρίτο πυλώνα η τραπεζική ενοποίηση που είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Και αυτός ο πυλώνας δεν προχωράει παρότι η, Κομισιόν έχει προτείνει μια πρόταση και ένα χρονοδιάγραμμα. Άκουσα και την κυρία Λαγκάρντ προχθές μετά το Eurogroup να υποστηρίζει θερμά αυτή την άποψη. Και τον κύριο Ντράγκη να υποστηρίζει ότι χωρίς τον Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Τραπεζικών Καταθέσεων δεν μπορεί να υπάρχει τραπεζική ενοποίηση και ισχυροποίηση απέναντι στους συστημικούς κινδύνους. Επειδή ορισμένα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο κρατάν καθυστέρηση και θέλουν να μην γίνει αυτό. Ποιο είναι το σχόλιο της Κομισιόν. Το δεύτερο, σημειώσατε ότι ε, η Ευρωζώνη υποφέρει από χαμηλές επενδύσεις, οι οποίες παραμένουν πολύ ε, χαμηλές σε σχέση με τις ανάγκες και σε σχέση με τα επίπεδα πρώτης κρίσης. Σε μια έκθεση που κάνατε ως Κομισιόν επισημάνατε ότι θα μπορούσε να, να υπάρξει μια πρόσθετη ενίσχυση των επενδύσεων ιδιαίτερα από τις χώρες με υψηλό εμπορικό πλεόνασμα, όπως είναι η Γερμανία, που υπερβαίνει τα όρια που προβλέπουν οι κανόνες. Ε, και επίση έχετε επισημάνει την ανάγκη να ενισχυθούν ιδιαίτερα οι επενδύσει και στις χώρες του Νότου. Θα ήθελα που έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά επενδύσεων σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο. Και γι' αυτό θα ήθελα την άποψή σας και τι πρωτοβουλία σκοπεύει να πάρει η Κομισιόν προς αυτή την κατεύθυνση. Uh, ε, okay. Δύο ερωτήσει λοιπόν για την πρώτη. Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Όντω, τον έφερα άλλωστε και στις αγωγικές μου παρατηρήσεις. Έχει τρεις πυλώνες τραπεζική ένωση. Ενία, εποπτεία και καθάριση έχουν ήδη προχωρήσει. Και το τρίτο, ο τρίτος πυλώνας αφορά το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Γι' αυτό και έχουμε προτείνει νομοθετική πρόταση σε αυτό το χρονικό σημείο το θέμα έχει περάσει στα χέρια των συνομοθετών, το Συμβούλιο δηλαδή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από εκεί θα περάσει για να προχωρήσει το θέμα αυτό. Βεβαίως παραμένουμε σε στενή επαφή και με τους δύο συνομοθέτες. Η δουλειά σε επίπεδο Συμβουλίου, παραδείγματι, έχει προχωρήσει στη συλλογή πληροφοριών για να εξασφαλιστεί η Συμβουλή των Τραπεζών προσαρμοσμένη στον κίνδυνο στο σύστημα αυτό με βάση τις αρχές ότι όποιος αναλαμβάνει πιστοκίνδυνο κίνδυνο θα πρέπει να συμβάλλει και περισσότερο στο σύστημα και επίσης παρακολουθούμε τις εργασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του κυρία Αστέρντε Λάγκε Άρα είναι στα χέρια των συνομοθετών η υπόθεση αυτή για να προχωρήσει. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε την υποστήριξη και, ό,τι μπορούμε, και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε τις εξέλιξεις αυτές. Για το δεύτερο θέμα, επενδύσεις. Για τις επενδύσεις υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, αξιόλογες, Κάποιες ε, από αυτές, τις οποίες αναφέρεστε, είναι νέες πρωτοβουλίες στο έγγραφο αναλογισμού επί παραδείγματι για την ενίσχυση και την εμβάθυνση της Νομισματικής Ένωσης. Αναφερόμαστε σε τρεις επιλογές για την ε, σταθεροποιητική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Και βασικά αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι είναι διαθέσιμες οι επενδύσεις. Είναι βέβαια πάντα η πρώτη δαπάνη που περικόπτεται σε περίπτωση κρίσης, αλλά ταυτόχρονα είναι αυτές οι οποίες αποτελούν και εγγύηση μέλλοντο για μια οικονομία. Άρα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να προσαρμόζουν τις επενδύσεις τους ή να τις τονώνουν, να τις ενισχύουν ακόμη και σε ε, οικονομικά δεινές εποχές. Αυτές είναι οι προτάσεις που θα περάσουν πλέον σε μια πιο συγκεκριμένη διατύπωση στο έγγραφο. Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Αττικές Επενδύσεις, Ερωτικά Ταμεία, διαθέσιμα στα κράτη-μέλη ή συγκεκριμένα για να μιλήσουμε για την Ελλάδα, ένα συγκεκριμένα στοχευμένο σχέδιο για την ανάπτυξη και τη εργασία στην Ελλάδα, προχωρούν και με έκτακτα μέτρα μάλιστα που εισάγουμε για να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Επομένως, ναι, οι επενδύσεις είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καταγράφονται και με πρακτικές δράσεις. Η Πρόεδρος, ξέρω ότι είναι πολλές οι ερωτήσεις, αλλά στο δυνατόν πιο σύντομα σας παρακαλώ να τις διατυπώνετε. Ο κύριος Γκίγκολτ, πράσινη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη πρόκληση που μου επιβάλλετε. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο όπως είπε και Νίνα γκίλ. Θέλω να σας καλωσορίσω και να υποστηρίξω και να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου για την ηγετική δράση που έχετε αναλάβει στην ενίσχυση των αγορών ε, και σας συγχαίρω για αυτά. Ωστόσο, έχω και λιγότερο ευχάριστα θέματα να εγείρω. Επί παραδείγματι, η υλοποίηση του BRRD στην περίπτωση του Επηρέας και την περίπτωση του Μπάνκο Popular συγκεκριμένα, καθάριση λοιπόν τραπεζών. Και νομίζω ότι εδώ δεν τρέχουμε τον κίνδυνο να ανατρέψουμε την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει κανείς στην Τραπεζική Ένωση. Οι διατάξεις της προληπτικής ανακεφαλοποίησης που προβλέπονται στην Περαραντή στηρίζονται και σε ε, ενάψματα που έχει δώσει η δική μας επιτροπή, ωστόσο έχουν παραμείνει αρκετά περιορισμένες. Η ανακεφαλαιοποίηση λοιπόν είναι πολύ περιορισμένη, σπάνια και υπό πολύ συγκεκριμένες ε, συνθήκες νομικά. Ερωτώ λοιπόν κύριε Επίτροπε, είστε διατεθειμένος να μας αποστείλετε γραπτός και λεπτομερός τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι στην περίπτωση του MPS της Μοντεπάσκη έχετε ε, θεωρήσει ότι πληρούνται όλοι οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης και επίσης μπορείτε να μας πείτε γιατί ενώ η περίπτωση της Μόντεντε Ιπάσκη έχει προχωρήσει τόσο καιρό πλέον βρισκόμαστε ακόμη σε αξιολόγηση, επίπεδο αξιολόγηση δεδομένων του 2014 χωρίς αξιολόγηση ενεργητικού που θα ε, εξασφάλιζε ε, την ε, επιβεβαίωση της βιωσιμότητας και της φερεγιότητας της τράπεζας. Επίσης, Στη Μόντε Πάσκη όλοι θα συμβάλλουν, θα λάβουν αποζημίωση ε, όλοι οι επενδυτές, Ανεξαρτούστον των είναι εκατομμυριούχοι, έχουν δηλαδή επενδύσει εκατομμύρια σε ομόλογα, πράγμα το οποίο θα οδηγούσε σε άνηση μεταχείριση σε σχέση με τους επενδυτές της Banco Popular που χάνουν την επένδυσή τους. Γιατί οι Ισπανοί επενδυτές βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους Ιταλούς. Απάντηση αρκετές ερωτήσεις σας. Στη σύγκριση Monte Dei και Μπάνκο Ποπολάρ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δύο τράπεζες είχαν ακολουθήσει διαφορετικές διαδικασίες και οι δύο με βάση τον BRRD στην περίπτωση της Monte Dei προληπτική ανακεφαλαιοποίηση στην περίπτωση Banco Popular εκαθάριση. Επομένως υπάρχουν διάφορες ε, προϋποθέσεις για την προληπτική ανακεφαλοποίηση. Καταρχάς δεν πρέπει να είναι σε πτώχευση ή σε κίνδυνο πτώχευση η τράπεζα. Είναι κάτι το οποίο και ο, ο μηχανισμός είναι αυτός, ο μηχανισμός θα προσδιορίσει. Και δεύτερον, οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν δεν θα καλυφθούν από κρατικές ενισχύσεις. Αυτές είναι λοιπόν οι προϋποθέσεις. με βάση τις οποίες έγινε και η προληπτική ανακεφαλοποίηση για την MPS, τη Μοντενταϊπάσκη, και ταυτόχρονα αυτό συνοδεύτηκε από ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της τράπεζας. ώστε να μπορέσει να επανέλθει σε βιωσιμότητα. Και όπως γίνεται και στην περίπτωση των κρατικών ενισχύσεων υπήρξε η υποχρέωση της συμμετοχής των επενδυτών και των μετόχων και μάλιστα στην περίπτωση των επενδυτών, λιανικής συγκεκριμένα, έγινε, δόθηκε αποζημίωση για τις κακές πωλήσει προς αυτούς. Η περίπτωση της Banco Popular ήταν διαφορετική. Γιατί ο SSM κατέληξε πως πτωχεύει ή είναι σε κίνδυνο πτωχευση η Banco Popular. Επομένως δεν χωρούσε πλέον ε, προληπτική ανακεφαλαιοποίηση. Και έτσι υπήρχε στο SRB η περίπτωση της τράπεζας που αποφάσισε την εξυγίανση. Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Αξιολόγηση του SSM, του Μηχανισμού Σταθερότητας, για τον κίνδυνο πτώχευσης. Για το EQR 2014 χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα δεδομένα και η Επιτροπή βεβαίως είναι έτοιμη να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις σας με τις απαραίτητες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Η ευθυντή τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είστε επίτροπο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αυξήσει το χρηματοπιστωτικό κίνδυνο, γιατί πρόσφατα προτείνατε την επανεγκατάσταση τη ε, καθάριση ευρώ εκτό Λονδίνου. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν μεγάλοι συστημικοί κίνδυνοι, 900 δις περίπου ευρώ κυρίω ε, σε παράγωγα ε, καθαρίζονται μέσω Λονδίνου. Αλλά η υποχρεωτική μετεγκατάσταση θα το κάνει πιο επικίνδυνο, πιο περίπλοκο και πιο δαπανηρό. Εσείς είπατε πως θα είναι το τελευταίο καταφύγιο. Αλλά ποιος και με πόση ειδοποίηση θα προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Οι επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στο παγκόσμιο σύστημα. Αλλά η δική σας πρόταση θα ε, διπλασιάσει πολλά κόστη. 77 δις ευρώ έχουν υπολογιστεί, που τελικά θα επιβαρύνουν τους πελάτες του συστήματος στην Ευρώπη. Το Λονδίνο έχει εκαθάριση σε γεν, σε γιοάν, σε δολάριο, σε αυστριλιανό δολάριο και παρόλα αυτά δεν είναι σε ένωση με καμία από αυτές τις χώρες και οι επενδυτές δεν έχουν πρόβλημα και δεν έχουν ζητήσει επαναγκατάσταση ούτε οι ίδιοι ούτε οι αρχές τους. Δεν ανησυχώ μόνο εγώ από αυτή την προστευτευτική, απομονωτική Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο Μάικλ Σπένσερ που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΝΕΚ που είπε πως εδώ μιλάμε για εθνικισμό που είναι τελείως κατά των ελεύθερων αγορών. Ο Σκοτ Ομάλε της ISDA είπε πως η επανακατάσταση και η απέτηση για αυτήν θα μπορούσε να έχει μαζικές συνέπειες για τις αποτελεσματικές διασυνοριακές ροές. Ο Τζιαν Κάρλο Κρίστοφερ από τις Ηνωμένες Πολιτείες είπε πως το να κάνουμε κάτι τέτοιο όπου ζητώντα αυτά τα νομίσματα να εκαθαρίζονται από συγκεκριμένε τοποθεσίε, σημαίνει πως θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο έκθεση στο άνοιγμα αυτό σε διάφορους συνελεγματικούς κινδύνους και θα γίνουν όλα πολύ πιο περίπλοκα. Άρα λοιπόν, αν προσπαθεί κανείς να ενισχύσει το ευρώ και την φήμη του παγκοσμίου, τότε η δική σας προστατευτική πρόταση είναι ένα βήμα πιστοχώρησης και φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το ευρώ ως ε, παγκόσμιο νόμισμα αποθεματικών. Γιατί θεωρείτε πως είναι τόσο εύθρα στη Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζεται να απειλεί με τέτοιου είδους χρηματοπιστωτικό γεωμπλοκάρισμα και δεύτερον, γιατί φοβάται τις αγορές τους πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί δεν αφήνει την επιλογή στους ε, καταναλωτές. δύο λεπτά όλοι σας παρακαλώ πολύ, όχι πάνω από δύο λεπτά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Επίτροπε. On, λοιπόν, ε, Για την πρόταση CCP έχω απαντήσει ήδη δύο φορές σχετικά με το σκεπτικό που διέπει αυτή την πρόταση Κομισιόν. Δεν έχω και πολλά δηλαδή να προσθέσω όσον αφορά τη λογική της πρότασής μας για το πώς ε, καταρτίστηκε, πώς, πώς αξιολογούμε τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους, πώς ε, βλέπουμε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις. Να έρθω όμως στα συγκεκριμένα θέματα που θέσατε. Πρώτον, ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις. Αυτά περιγράφονται με ακρίβεια στην νομοθετική μας πρόταση, η ΕΣΜΑ και η ΕΚΤ, που θα διαβολεύονται και με τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και στη συνέχεια η Κομισιόν λαμβάνει απόφαση βάσει των προτάσεων που θα τις υποβάλουν αυτές οι αρχές. Δεύτερον, ακούστηκαν διάφορα στοιχεία όσον αφορά τον αντίκτυπο. Είπατε ότι μπορεί μέχρι και να διαπλασιαστεί το κόστος. Η μελέτη αντικτύπου μας δείχνει ε, μια αύξηση των περιθωρέων κατά 8 έως 12%. Ούτε εδώ εισάγουμε μια πολιτική με βάση τον γεωγραφικό χώρο γενικά. Είναι όμως μία από τις επιλογές που έχουν η ΕΣΜΑ και η ΕΚΤ σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι ασφαλιστικές δικλείδες και δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, η συγκέντρωση δημιουργεί και αυτή ορισμένους κινδύνους τους οποίους θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Να πω ότι τα, η εκαθάριση παραγόγων ε, που είναι ε, ε, εκπεφρασμένα σε γεν διέπεται από γεωγραφική πολιτική. Για το ENF, ο κύριος Άνεμανς. Το είπα καλά. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Αν δεν σας πειράζει. Στο τελευταίο ερώτημα του κύριου Κόμπερν. Μιλήσατε για την ε, αναθεώρηση της ε, Ένωσης κεφαλαιογορών, Όπως είδαμε το Brexit είναι να εξελίξη. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει αυτό. Η αρχή της εναρμόνισης πώς θα εφαρμοστεί. Γενικά ή εξειδικευμένα. Είναι 551.000 οι εργαζόμενοι στο χρηματοπιστωτικό τομέα. 80 δισεκατομμύρια είναι ο όγκος των συναλλαγών του. Όλοι ξέρουν ότι θα οδηγηθούμε σε μια απώλεια αποτελεσματικότητας, απώλεια ρευστότητα, Γιατί λοιπόν δεν φροντίζεται για ε, ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα ε, να μην ε, σπέβδει με μεγάλη σπουδή η κεφάλαια αγορά, αλλά να προσαρμοστούν οι ρυθμοί τους. Γιατί λοιπόν πατάτε τον γκάζι αντί να προσπαθείτε να επιβραδύνετε. Ε, well, ε, on, Brexit. Για το Brexit και τι επραγματεύσεις του Brexit. Όπως ξέρετε, Ξεκίνησαν μόλις εχθές η διαπραγματεύση για τον Brexit. Ένα πρώτο σύνολο θεμάτων που αφορεί, αφορά τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ε, σύνορα μέσα στην ίσο της Ιρλανδίας, και τι είναι οι προτεραιότητες και οι μελλοντικέ βέβαια ε, ε, για τα λοιπά θέματα του Brexit ε, θα προχωρήσουν όταν έχουν κλείσει τα τρία αυτά πρώτα θέματα. Πάντως, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται ακόμα να εξετάσουμε και να μας απασχολήσει στο τι θα γίνει όταν η μεγαλύτερη κεφαλαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγει εκτός της Ένωσης. Και κάθε υπόθεση βέβαια θα αναπτυχθεί με βάση αυτό το δεδομένο. Όταν το γεγονός ότι η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά βγει έξω από το πλαίσιο της ΕΜΙΡ, το πλαίσιο δηλαδή του κανονισμού για τις ευρωπαϊκές κεφαλαίες Αγόρε, τότε θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε στο γεγονός αυτό και αυτό είναι, κομμάτι της, αυτό είναι ο λόγος μάλλον για τον οποίο αποβάλλουμε την πρόταση που καταθέσαμε. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκό Λαϊκό. Όχι, έχω ακόμα δύο λεπτά, Πρόεδρε. Διότι, αν καταλαβαίνω καλά, δεν αποκλείεται εσείς στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Brexit να γίνει προσπάθεια για ανάπτυξη νέων σχέσεων με το Λονδίνο και όχι να θεωρηθεί το Λονδίνο απλώς ως ε, μια αγορά έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αφήνεται ανοιχτό το παράθυρο ή την πόρτα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα μπορούσε το Λονδίνο ως χρηματοοικονομικό κέντρο να διατηρήσει στενές, στενούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε μια ευέλικτη ε, αντίληψη και όχι μια αντίληψη που απλώς ξεφορτώνεται ούτως επί το Λονδίνο. Κύριο Ναπρόφσκης. Να σας απαντήσω. Η πρόταση, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, είναι μια πρόταση που δεν είναι συγκεκριμένα μόνο για ένα κράτος. Δηλαδή, είναι μια πρόταση που αφορά τις τρίτες χώρες και τα, τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους εκεί και βέβαια αυτό μπορεί να έχει και κάποιες συνέπειες και για κεντρικούς αντισυμβαλόμενους πέραν του Ηνωμένου Βασιλείου. Οπότε, μην το αντιμετωπίζετε περιοριστικά ως μια πρόταση που έχει να κάνει μόνο με ένα κράτος μέλος. Και πάλι, ε, θα επαναλάβω πως εξήγησα το σκεπτικό με το οποίο υποβάλαμε την πρόταση αυτή, η οποία αυτή τη στιγμή έχει πάει στους νομοθέτες και νομίζω το κοιτάει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Και Χόκμαρκ, σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για τις ε, αναθεωρήσεις που έχετε κάνει για την ιεράρχηση κτλ. Νομίζω πως ε, και στο δικό μου κείμενο θα διατυπώσω για το θέμα της ιεράρχησης, κάτι αντίστοιχο και θα πω στην Επιτροπή να το κάνουμε με διαδικασία fast track για να μπούμε και στους ίδιους ρυθμούς με τους υπολείπους. Για την παρουσίαση που μας κάνατε προηγουμένως, θέλω να επανέλθω στην Ένωση Κεφαλαιογορών. Γιατί αυτή τη στιγμή τρέχει κάτι το πολύ μεγάλο και βέβαια έχει να κάνει και με τις διαπραγματεύσεις με τον Brexit. Οπότε θα ήταν ενδιαφέρον για μας να μας πείτε εσείς πώς θεωρείτε πως θα επηρεάσει το Brexit τις ευκαιρίες ε, δημιουργίας μιας ισχυρής ένωσης Και επίσης, χρηματοπιστική σταθερότητα και κίνδυνη ε, επειδή το σύστημα θα διαιρεθεί και το city είναι μεγάλο. Έχει ένα τέτοιο μέγεθος που δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί πως μπορούμε να έχουμε μια κεφαλογορά σαν αυτή που έχουμε σχεδιάσει προ-Brexit. Οπότε αν μπορείτε εδώ να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη διευκρίνηση για το τι θα γίνει με την ιεράρχηση των πιστωτών. Αυτό είναι εξαιρετικά ε, καλοδεχούμενο και το Συμβούλιο το πακέτο το έχει συμφωνήσει. Οπότε και εκεί θα ακολουθήσει μια διαδικασία φαστρά Αν το κάνει και το Κοινοβούλιο, νομίζω ότι αυτό ε, μας οδηγεί στο να κλείσουμε τη δουλειά αυτή φέτος. Και μετά αυτό θα μας επιτρέψει οι τράπεζες να οικοδομήσουν αυτές τις ε, επαρκείς ζώνες απομόνησης, αυτά τα buffer, μέσα στον κατάλληλο χρόνο. Τώρα, για να έρθω στο θέμα του Brexit και του πώς θα επηρεάσει αυτό ε, την ε, Ένωση Κεφαλαιογορών και τα όσα μόλις περιγράψατε, να σας πω πως το Brexit θα κάνει πιο προκλητική την προσπάθεια να δημιουργήσουμε αυτή την αγορά ε, την Ένωση Κεφαλαιογορών αλλά ξέρετε, θα γίνει και πιο σημαντικό. Γιατί βέβαια θα έχουμε τις κεφαλογορές και στα 27 κράτη-μέλη που θα ενισχυθούν και θα το δούμε αυτό στην ενδιάμεση αναθεώρηση όπου θα διαπιστώσετε πως γινόμαστε πιο φιλόδοξοι Θέλουμε να καταθέσουμε νέες προτάσεις, νέες ιδέες σχετικά σε αρκετά σημεία. Εν πάση περιπτώσει ο στόχος μας είναι να μειώσουμε τα εμπόδια στην Ευρώπη ώστε να έχουμε μια κλιμάκωση και μεγένθηση των εταιριών με καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση διασυνοριακά και με πλήρη χρήση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς που αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται στις πλήρεις δυνατότητες που έχει. Ευχαριστώ. Έχετε λίγο χρόνο αν θέλετε να επανέλθετε. Χωρίς να είναι αναγκαίο βέβαια. Ευχαριστώ. Σοσιαλιστές ο κύριος Σάντ. Δύο ερωτήματα. Το πρώτο σχετίζεται με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που είναι ένας ε, τομέας που διευρύνεται ταχύτατα και που ενισχύει και τις οικονομίες των περιφερειακών κράτων μελών. Ωστόσο, επλήγησαν οι υπηρεσίες αυτές ε, από τα πρόσφατα σκάνδαλα. Μάλιστα βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ε, γύρω από τα ζητήματα της φοροποφυγής, φοροδιαφυγής ε, και τα λοιπά. Και ο ανταγωνισμός ε, στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα γίνει ακόμα πιο αδυσόπιτο στα επόμενα χρόνια. Τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική. Οι πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να παραμείνουν σε εξαιρετική κατάσταση ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της Ένωσης Κεφαλαιογορών. Πρέπει να ε, αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις από, τις, από τους πολιτικούς και από, τα, από τους δημοσιογράφους. Ε, μήπως θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή πρόβλεψη ε, μήπως δεν θα, θα πρέπει να υπάρχει αυτορύθμιση αλλά να τεθεί επικεφαλής μια δημόσια αρχή προκειμένου να εξασφαλίζει τη διαφάνεια. Δεύτερον, όσον αφορά το τομέα των ασφαλίσεων. Η οδηγία για την αναδιανομή των ε, ασφαλίσεων θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο έως το 2018. Υπάρχουν τέσσερις εκτελεστικές πράξεις που αφορούν τη διακυβέρνηση, την εποπτεία των προϊόντων, καθώς και την αξιολόγηση της καταλληλότητας της υποβολής εκθέσεων. Οι εκτελεστικές πράξεις είναι δεσμευτικές για τα κράτη-μέλη που πρέπει να τις εφαρμόσουν έως τις 23 Φεβρουαρίου 2018 με σοβαρές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις. Μιας και η Κομισιόν δεν έχει ακόμη εκδώσει ε, τις ε, εκτελεστικές αυτές πράξεις, αναμένεται αυτό να γίνει μόλις τον Οκτώβριο και έτσι μένει πολύ λίγος χρόνος στα κράτη-μέλη. Και έτσι θα πληγούν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι ρεαλιστικός ο χρόνος εφαρμογής όλων αυτών και αντίκειται η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην αρχή της αναλογικότητας. Στη χώρα μου οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές ή μικρομεσαίες και έτσι θα ε, κληθούν να υπομισθούν ένα δυσανάλογο ε, άχθος. Θα μπορούσε η Κομισιόν να εξετάσει ενδεχόμενο αναβολή της εφαρμογής της θέσης ισχύω της οδηγίας IDD. Ευχαριστώ. Πάλι δύο ερωτήματα μου θέσατε. Το ένα αφορά τις χρηματοδοτικές υπηρεσίες και το άλλο αφορά την, ε, και την ε, φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή και το άλλο αφορούσε τα IDD. Να ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα. Υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί Αναφερθήκατε κι εσείς σε κάποιους ε, στον τομέα της φορολογίας, όπου εφαρμόζουμε την πρωτοβουλία του ΟΣΑ για την καταπολέμηση της, ε, μεταβίβασης των, των, ε, της εσωτερικής μεταβίβασης των κερδών και αυτά που αποφασίστηκαν σε επίπεδο ΟΣΑ εφαρμόζονται και εδώ στην Ευρώπη και μάλιστα με μια ακόμη πιο φιλόδοξη ατζέντα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ενισχύουμε τους κανόνες μας για την ε, καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, βρώμικου χρήματος. Ε, η οικονομική σύμβουλη, η ενδιάμεση, υπόκεινται ήδη στους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων βάσει αυτής της οδηγίας και σχεδιάζουμε και περαιτέρω βήματα για την ενίσχυση της ευθύνης ε, την οποία επομίζονται οι σύμβουλοι και η ενδιάμεση για, για τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Και η πρόταση αυτή θα δημοσιευθεί πολύ σύντομα. Άρα, επί της ουσίας, λοιπόν, έχουμε σκοπό να αναλάβουμε μια σχετική νομοθετική πρόταση να υποβάλουμε μια σχετική νομοθετική πρόταση για την αντιμετώπιση ε, εκείνων που προβαίνουν σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και αξιοποιούν τυχόν νομοθετικά κενά. Και ε, στο πλαίσιο αυτό υπάρχει και η πρόταση για την υποβολή εκθέσεων αναχώρα, αλλά και η οδηγία για την καταπολέμηση της ε, νομιμοποίησης παράνομων Υπάρχει δηλαδή ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι μεγάλο έργο, ε, αφορά και, την, και το πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση, το οποίο επίσης προσφέρει ως μέσα ασφαλιστικές δικλείδες. Και βεβαίως μπορούμε να δούμε ε, και περαιτέρω τρόπους για την ενίσχυση. Στο δεύτερο ερώτημά σας. Όσον αφορά την εφαρμογή τι οδηγίες για την αναδρομή των ασφαλίσεων, οι εκτελεστικές πράξεις που θα εγκριθούν βάσει της IDD θα πρέπει να είναι πλήρως συμπατές με την οδηγία, όπως θα ε, υιοθετηθούν από τους συνομοθέτες, θα μπορούν να ε, ορίζουν συγκεκριμένες ε, λεπτομέρειες αλλά όχι να αναθεωρούν το πνεύμα της, της οδηγίας και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο κατάρτισης αυτών των εκτελεστικών ε, ε, πράξεων βάσει των συστάσεων που έχουμε λάβει από την ΕΙΟΠΑ. Οι διαδικασίες αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη και θα εγκριθούν οι εκτελεστικές αυτές τις πράξεις τις επόμενες εβδομάδες σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη προκειμένου να διευκολύνουμε τα κράτη-μέλη και στη διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Ε, στην ουσία δηλαδή προσπαθούμε να ε, εγκρίνουμε και να δημοσιεύσουμε αυτές τις εκτελεστικές πράξεις το συντομότερο δυνατό ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν ωστόσο ε, θα ήταν λάθος να αναβάλουμε την θέση σε ισχύ της IDD υπήρξε μια απόφαση για περίοδο χάριτος δύο ετών και πρέπει να γίνει σεβαστή η περίοδος χάριτος αυτή ε, γιατί ε, ήταν επαρκές ε, το χρονικό αυτό διάστημα. Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία τόσο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και με τα, με το, με τα κράτη-μέλη προκειμένου να δοθεί η, απαραίτητη ασφάλεια δικαίου σε όλους τους εμπλικόμενους φορείς. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Έχουμε άλλα 10 λεπτά για το θέμα αυτό και έχουμε τέσσερις ομιλητές. Παρακαλώ λοιπόν ε, να τηρήσετε ε, το όριο των δύο λεπτών και λιγότερα θέματα παρακαλώ, αν, αν, μπορείτε. Ε, εσύ το έκανες. Για να δούμε, κύριε Κίρτσο, θα τα καταφέρετε. Δύο ερωτήματα. Η κυβέρνηση των ΙΠΑ προχωρεί σε απορρίθμιση του τραπεζικού τομέα. Εσείς κύριε Πίτροπε, πώς πιστεύετε πρέπει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εμείς ε, χρειαζόμαστε με έναν σταθερό τραπεζικό κλάδο, αλλά πρέπει αυτός ο κλάδος να είναι και ανταγωνιστικός στην παγκόσμια αγορά. Πρόκειται δηλαδή για μια πρόκληση που μας θέτει η ΕΠΑ. Δεύτερο, ε, ερώτημα αφορά τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα. Η κατάστασή του κατά τη γνώμη μου βελτιώνεται, αλλά αργά και χρειαζόμαστε έναν πιο δυναμικό τραπεζικό κλάδο προκειμένου να μπορέσει να αναπτυχθεί η οικονομία. Η Κομισιόν έχει προτάσεις ή ιδέες, ε, θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία προκειμένου να επιταχυνθούν ε, τα θετικά σημάδια που δείχνει ε, το τελευταίο διάστημα ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές και να σας πω καταρχήν Ποιες είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για τη ΣΥΠΑ. Για την αναθεώρηση Dodd Frank. Ξέρετε πως πρόσφατα δημοσιεύθηκε ένα νομοθέτημα το οποίο αυτή τη στιγμή εμείς αξιολογούμε και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις εκεί. Βεβαίως, το μήνυμα που στέλνουμε στις αρχές της ΕΠΑ είναι πως αναμένουμε μια συνεχιζόμενη ε, συμμόρφωση με τα διεθνή ε, πρότυπα και κανόνες, για παράδειγμα αυτούς της Βασιλείας, για την χρηματοδότηση, για το χαρτοφυλάκιο κτλ. Κομμάτια δηλαδή τα οποία βρίσκονται και στο δικό μας ε, πακέτο για τις τράπεζες που παρουσιάσαμε τον Νοέμβριο και βεβαίως θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα βήματα που χρειάζονται στην πράξη, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για συστάσεις και θα πρέπει να δούμε τι είδου συνέχεια θα δοθεί από, την, ε, από τις αρχές των ΙΠΑ, από το Κογκρέσο και από τη Γερουσία. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ε, τι θα συμβεί ακριβώς και ποιες θα είναι οι εξελίξεις με την αναθεώρηση Dodd Frank δεν έχουμε πρόβλημα με την ίδια αναθεώρηση. Και εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε αναθεώρηση της δικής μας νομοθεσίας με την αναλογικότητα, με στοχευμένες προσαρμογές. Αλλά δεν θα πρέπει αυτή η αναθεώρηση να σημαίνει απορρίθμιση και δεν θα πρέπει να σημαίνει απομάκρυνση από διεθνώς ε, συμφωνημένα πρότυπα. Τώρα για τη δεύτερη ερώτηση που κάνατε, για τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, και θα συμπεριλάβω εδώ το θέμα των κόκκινων δανείων και το ποσοστό των μη εξυπηρετώμενων αυτών δανείων, έχει αναφερθεί πως αυτό αποτελεί κομμάτι του ε, προγράμματος στήριξης της Ελλάδος. Γιατί εκεί είχαν διατεθεί κάποιοι πόροι για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, γιατί αντιμετώπιζε ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα προβλήματα. Και βεβαίως παρακολουθούμε πολύ στενά και εκεί τις εξελίξεις. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι πως υπάρχει ανάγκη για στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα με ευρύτερους όρους και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε καταθέσει αυτό το σχέδιο για θέσει εργασίας και ανάπτυξη στην Ελλάδα που συμφωνήθηκε το 2015 ε, όταν ξεκίνησε να τρέχει το ε, μνημόνιο στην Ελλάδα. Και την περασμένη εβδομάδα παρουσιάσαμε και κάποια αξιολόγηση για το τι έχει συμβεί ε, τα τελευταία δύο χρόνια και πόση στήριξη έχει κινητοποιηθεί προς την Ελλάδα μέσω του σχεδίου αυτού, δηλαδή διευκόλυνση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τεχνική βοήθεια όπως επίσης και μπροστοβαρής χρηματοδότηση, έτσι ώστε η Ελλάδα να μην έχει πρόβλημα ρευστότητα στη στιγμή της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων ε, και επίσης μέσω του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου επιπλέον χρηματοδότηση και άλλων μεσών, έτσι ώστε το σχέδιο αυτό για την ανάκαμψη, την ανάπτυξη, με συγχωρείτε, και τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα να προχωρήσει. Είναι ο κοινό μας στόχος άλλωστε, η ελληνική οικονομία να ανακάμψει και με επιτυχία να κλείσει το ε, πρόγραμμα βοήθειας, το πρόγραμμα διάσωσης και να μπορέσει να επιστρέψει στις αγορές η Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Από τους ε, σοσιαλιστές ο κύριος Βέτσακερ. Σάκερ. Θα συνεχίσω με τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους και για ένα θέμα το οποίο έχει ακολουθεί έχει συζητηθεί πολύ επανεγκατάσταση. Να σας συγχαρώ, να σας συγχαρώ για τις προτάσεις σας. Καλό είναι αυτή η προσέγγιση που βασίζεται στην επικινδυνότητα και δεν προδικάζει το αποτέλεσμα, αλλά λέει τι συμβαίνει, κλασικό σχήμα τρίτης χώρας ή ε, με υποπτία ή ε, πολιτική με τόπο εγκατάστασης. Όλα αυτά θα αποφασιστούν όταν υπολογιστούν οι κίνδυνοι κάθε εναλλακτικού σενάριου. Και επίσης να σας συγχαρώ από το συλλογικό υποπτικό όργανο σε μία πιο ενιαία ε, ε, εποπτική υποπτική αρχή για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους, χωρίς όμως βέβαια να έχετε φτάσει μέχρι το τέλος αυτός της διαδρομής, οπότε αυτό έχει πλεονεκτήματα και για τις εξωτερικές μας σχέσεις, αλλά και για τα εσωτερικά προβλήματα και για τη σύγχυση και για την περιπλοκότητα. Οπότε, πείτε μου, γιατί δεν πήγατε ένα βήμα παρακάτω, έτσι ώστε οι βασικοί κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι να έχουν μια ενιαία εποπτική αρχή, έσμα και ε, μηχανισμός ε, σταθερότητας που θα αποφασίζουν και ως αντίβαρο εάν θέλετε να έχετε την εποπτεία και την εκαθάριση, να κάνετε αυτό το οποίο ζητάμε η κυρία Σουίνμπορν και εγώ, για να δούμε αν μπορούμε να περάσουμε και ένα σύστημα με μια ενιαία αρχή εκαθάρισης που κάποτε είχε προταθεί. Θέλω να μου πείτε αν το ξανασκέφτεστε. Ναι. Για αυτές σας τις ερωτήσεις. Πρώτον, συνοδευτικές προτάσεις. Ενίσχυση της εντολής της συναλλαγέ στις συναλλαγές με κεντρικούς αντισυμβαλωμένους από τρίτες χώρες. Υπάρχει βεβαίως πρόταση. Και είναι, πιστεύουμε, ένα σημαντικό βήμα στην εποπτεία να είναι σαφής ποιος είναι ο κεντρικός αντισυμβαλόμενος για την ευρωπαϊκή πλευρά, για να υπάρχει συνεργασία με τις αρχές των τρίτων κρατών και να υπάρχει αυτή η δίκτυ εποπτεία. Σε αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε την εντολή της ΕΣΜΑ. Επίσης αναφερθήκατε στην εντολή της ΕΣΜΑ και εσωτερικά, στην ενίσχυση της εσωτερικά. Όντως, προχωρούμε σε αναθεώρηση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών που θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο. Προς το παρόν έχουμε ολοκληρώσει τη δημόσια διαβούλευση με 220 απαντήσεις που κατατέθηκαν από του εμπλεκόμενου φορείς και ένας από του στόχου μας είναι η ενίσχυση της ε, κεντρικού χαρακτήρα λήψη αποφάσεων για την εποπτεία, για όλες τις εποπτικές αρχές, περιλαμβανομένες και τις ΕΣΜΑ. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουμε την ΕΣΜΑ στην αναθεώρηση. έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και την εποπτική σύγκληση που χρειάζεται για την ομοιόμορφη υλοποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων, άρα και των εποπτικών δραστηριοτήτων και πρακτικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι πως οι κανόνες εφαρμόζονται παντού με τον ίδιο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν υπάρχει ότι δεν γίνονται κάπου εκπτώσεις ως προς την ε, λιγότερο αυστηρή τήρηση των όρων προκειμένου να προσελκυστούν ορισμένου τύπου δραστηριότητες επιχειρηματικές. Ε, για την άλλη σας ερώτηση Γιατί δεν προχωρούμε κατευθείαν σε μία ενιαία εποπτική αρχή. Υπάρχουν κάποιοι παραγόντες που περιορίζουν τις δυνατότητες δράσης μας, πρέπει να τους λάβουμε, υπόψη. Αν και μακροπρόθεσμα θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και σκέψη. Καταρχάς έχουμε τις εθνικές δημοσιονομικές ευθύνες και αρμοδιότητες που, σημαίνει, ε, που σημαίνουν ότι ορισμένα κράτη-μέλη είναι επιφυλακτικά ως προς την διάθεση της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων που μπορεί να έχει δημοσιονομικές συνέπειε για ορισμένα σε ε, φορείς εκτός αυτών των ίδιων των κρατών μελών ή εκτός του ελέγχου των κρατών μελών. Άλλωστε παραδοσιακά έχουν ε, σαφή δράση οι εθνικές αρχές ελέγχου σε αυτές τις και δεν μπορεί να αλλάξει αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά πάντως πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των, των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και να προχωρήσουμε προς μια εποπτική σύγκληση. Ο κύριος Μπάλτς, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σε σχέση με την Banco Popular και την αναθεώρηση της ε, ΕΑΤ και βέβαια σε σχέση με την BRD χθε μας είπε η κυρία Νουή ότι η κρίση της Ισπανικής Banco Popular που οδήγησε στην εγκαθάριση της 7 ε, Ιουνίου δείχνει ότι χρειάζεται η εποπτική αρχή περισσότερες εξουσίες σε σχέση με τις αδύναμες πιστώσεις και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Συμφωνείτε σε αυτό και μπορούμε να περιμένουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδιώξει αυτή την κατεύθυνση με τις προτάσεις που θα κατατεθούν στο μέλλον. Δεύτερον, ένα άλλο χαρακτηριστικό της κρίσης ε, της Banco Popular λέγεται ότι γέννησε αμφιβολία σε σχέση με την ποιότητα των τεστ αντοχής. Πώς μπορεί δηλαδή να έχει ε, περάσει ένα τεστ αντοχής, τα τεστ αντοχής η τράπεζα αυτή και στη συνέχεια να κηρυχθεί σε πτώχευση, σε κίνδυνο πτώχευση, χωρίς να έχει ενδεχομένως αξιολογηθεί ένα σενάριο αντίξων εξελίξεων. Πώς γίνεται να ξέφυγε κάτι τέτοιο. Για τον κανονισμό, για την οδηγία για την κεφαλαία, για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Ο ΚΑ. Η κυρία Νουιέλα και η κυρία Λάουτσλέγκερ ενημέρωσαν την Επιτροπή από ό,τι μας είπαν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στα ε, τήσια μέτρα παρέμβασης στο πλαίσιο της ΟΚΑ και ότι σε αυτό κάνουν τις προτάσεις τους. Δεν ήταν πολύ σαφή τα πράγματα. Σε σχέση με την BRD, τα... το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονό ότι τα μέτρα είναι είτε πρόημα είτε όψιμα. Η Επιτροπή πώς το αξιολογεί αυτό που μας είπαν. Ευχαριστώ και για αυτές τις ερωτήσεις. Γιατί μην εξυπηρετούμε εξυπηρετούμενα δάνεια για την πρώτη σας ερώτηση. Βεβαίως είναι πιο γενικό το ερώτημα και όταν εξετάζουμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, πάνω απ' όλα θα δώσουμε έμφαση στην ε, ευρωπαϊκή εποπτική δράση και αυτό θα μας απασχολήσει στις συνομιλίες ε, του ΕΚΟΦΗΝ ε, του προσεχούς μήνα με το πρόγραμμα δράσης. Για να μιλήσω πιο συγκεκριμένα τώρα όπως είπα και στις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις, μετά από αυτή την πρώτη περίπτωση ε, καθάρισης τράπεζας, θα δούμε η της τράπεζα, θα δούμε ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες, τι περαιτέρω βήματα χρειάζονται και τι είδους μελήματα μένουν προς διευκρίνηση προκειμένου να, να ακολουθηθούν μάλλον οι προτάσεις ε, του μηχανισμού σταθεροποίησης. Μετά την εξυγένση θα τα αξιολογήσουμε όλα αυτά. Σε αυτό το στάδιο δηλαδή. Τώρα για τα τεστ αντοχής δεν μπορώ να κάνω σχόλια εκτεταμένα διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τραπεζική εποπτεία. Σημειώνουμε πάντως ότι η Banco Popular ήταν η τρίτη χειρότερη του τεστ αντοχής του 2016. Και από ό,τι γνωρίζω, κυρία Νουή σας είπε χθε ποια μέτρα είχε αναλάβει με αυτοψίες και με ε, ανακεφαλοποίηση. Για την ε, πρώιμη παρέμβαση. Ο στόχος της ε, πρώιμης παρέμβασης, της έγκυρης παρέμβασης, είναι η σταθεροποίηση μιας τράπεζας σε δυσκολία για να αποφευχθεί η εκαθάριση ή η εξυγίανση. Αυτό είναι συνήθις ε, και φυσιολογική δράση μιας εποπτικής δραστηριότητας με εξουσίες έγκαιρης παρέμβασης που προβλέπονται ήδη από το, Ευρωπαϊκό ε, Κανονιστικό Πλέγμα. Επομένως και με τον μηχανισμό και με το SRB εξετάζουμε πώς μπορούν να βελτιωθούν αυτοί οι κανόνες. Ευχαριστώ. Κύριος Πολ Τάν, Σοσιαλιστής Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δεπρόσωπο που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. CMU έχει ξεκινήσει και βρισκόμαστε στην φάση της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Κοιτάμε πώς μπορούμε να την καταστήσουμε πιο βιώσιμη, την Ένωση Κεφαλογορών. Το βλέπω και το θετικό είναι ότι η Κομισιόν με την ομάδα υψηλού επίπεδου της εργάζεται σκληρά ε, για την ενίσχυση της Ένωσης Κεφαλαγορών. Παρ' όλα αυτά, κάποιες φορές προσπαθώ ακόμη να καταλάβω ποια είναι συγκεκριμένα η πρόοδος που κάνει η Κομισιόν και ποια μπορεί να κάνει. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε κατευθυντήρες ε, γραμμές από την ΕΣΜΑ για την αρχή ESG. Επίσης έχουμε ε, συστάσεις από την Task Force γιατί τη χρηματοδοτήση θα, θα τις υιοθετήσει και η Κομισιόν και θα τις προωθήσει και στο G20 για να μπορέσουν να γίνουν και επιχειρησιακά να μπορέσουν να, λειτουργήσουν και στην πράξη αυτές οι, οι συστάσεις. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε την πρόταση για τις ε, ιδιωτικές συντάξεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει ε, καθορίσει τη δική του στάση ως προς αυτά τα ιδιωτικά, τις ιδιωτικές συντάξεις και είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο προκειμένου η Ένωση Κεφαλαιογορών να καταστεί πιο βιώσιμη. Ευχαριστώ. για το έργο αυτό ώστε να καταστεί η Ένωση πιο βιώσιμη. Είναι πράγματι μια από τις προτεραιότητες μας που επισημαίνεται και στην ανεδιάμεσα αναθεώρηση της Ένωσης Κεφαλαιογορών και ε, είναι και ένα θέμα που απασχολεί την, ε, ε, θα απασχολήσει την ομάδα υψηλού επίπεδου το πρώτο τρίμηνο του 2018. Θα γίνει όμως και μέσα στον ε, Ιούλιο μια, ένα συνέδριο ε, υψηλού επίπεδου για να συζητηθούν τα μέχρι στιγμής ευρήματα και πορίσματα. Όσον αφορά τις κατευθύνσεις γραμμές σχετικά με το ESG, και τα χρηματοπιστωτικά θέματα δεν υπάρχει ε, ορισμός αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ε, πίστη. Ωστόσο υπάρχουν διατάξεις ε, διάσπαρτες στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Και στην ενδιάμεσα αναθεώρηση θα ανακοινώσουμε και την πρόθεσή μας να εξετάσουμε αυτήν την, την υποχρέωση πίστης των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και την υποχρέωσή τους να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις διαστάσεις κατά τη λήψη αποφάσεων. Για την Task Force FSB για τις ε, πληροφορίες που σχετίζονται με το κλίμα. Έχουμε εξετάσει αυτές τις προτάσεις και τις έχουμε λάβει υπόψη μας στην, ε, στην, ε, στις επόμενες μα, γραμμές μας που είναι και ο, ο λόγος για τον οποίο αναβλήθηκε ε, για κάποιο χρονικό διάστημα η δημοσίευση τους ακριβώς για να μπορέσουμε στο μέτρο του δυνατού να λάβουμε υπόψη μας τις συστάσεις του FSB. Όσον αφορά αυτά τα πανευρωπαϊκά προϊόντα ιδιωτικών συντάξεων. Σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε τη σχετική μας πρόταση πριν από το καλοκαίρι. Και στην ουσία θα συμπεριλάβουμε την δυνατότητα να συνυπολογίζονται και παράγοντες ESG. Ε, χρειάζονται, χρειάζεται ένας ε, ε, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη αυτές οι διαστάσεις ε, στην, ε, στην ε, προ, διαδικασία κατάρρισης αυτής της νομοθεσίας. ένα λεπτό ο κύριος Αργιανόπουλος. Ε, ε, κύριε Ντομπρόσκη, πριν ε, από λίγο μιλήσατε για την Ελλάδα και για τη βοήθεια που δώσετε στις τράπεζες. Μιλάμε βέβαια για τα μνημόνια, τα οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός, και για την ανάπτυξη. Επικαλούμενη λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μια συζήτηση για το χρέος, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και την χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική σταθερότητα καταλήξατε πριν από λίγο σε ένα τέταρτο μνημόνιο που βέβαια δεν ψηφίζουν τα άλλα κόμματα αλλά υπόσχονται να το υλοποιήσουν και για σταθερότητα. Σταθερότητα ξέρετε τι σημαίνει κατά την άποψή σα. Σημαίνει πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2022 και μέχρι το 2060 2% για 37 χρόνια. Σημαίνει νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων για 16η φορά. Σημαίνει μισού των 250 ευρώ και τρομακτική φορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων με φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές στις μεγάλες επιχειρήσεις σημαίνει τη βέλτιστη πρακτική των ομαδικών απολύσεων που σήμερα στην Ελλάδα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σήμερα σημαίνει 15.000 απολύσεις συμβασιούχων στους Δήμους. Σήμερα. Τι μπορεί να περιμένει λοιπόν ο εργαζόμενο ή ο λαό τη χώρα μα από την πολιτική την οποία, την οποία τα σκήνηση μαζί με την ελληνική κυβέρνηση. Uh, well, uh, first of... Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που αξίζει να κάνουμε είναι να εξηγήσουμε το τρίτο πρόγραμμα στήριξης ποιο στόχο έχει. Έχει σκοπό να επανέλθει η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα και να εξασφαλίσουμε πως η ελληνική οικονομία ανακάμπτει. Και όντως, αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο βλέπουμε. Οι προβλέψεις μας θεωρούν πως θα έχουμε μία ανάπτυξη της τάξης του 2,1% φέτος και μία ανάπτυξη η οποία θα ξεπεράσει τις προβλέψεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν έχουμε την οικονομία που ανακάμπτει, την ανεργία που μειώνεται την χρηματοσφαιρική σταθερότητα που έχει επανέλθει και είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να μείνουμε σε αυτή την τροχιά. Αυτό που είπατε, εντάξει, είχαμε μία επιτυχή δεύτερη αξιολόγηση και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πληρωθεί η επόμενη δόση έτσι ώστε να καλύψει τις τρέχουσες χρηματοδοτικές ανάγκες και παράλληλα να προετοιμάσει την Ελλάδα για να επανέλθει στις αγορές έτσι ώστε η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της και να μην εξαρτάται από την οικονομική στήριξη και τα σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ κύριε Αντιπρόεδρε για το χρόνο που μας διαθέσατε. Ήσασταν πάρα πολύ υπομονητικός με τις επιπλέον ερωτήσεις. Νομίζω λοιπόν πως πρέπει να σας ευχαριστήσω. Γεια σας. Θα περάσουμε εμείς τώρα πολύ γρήγορα έτσι ώστε να κερδίσουμε χρόνο στο επόμενο σημείο της επόμενης ε, ε, το επόμενο σημείο τη ημερήσια κατά πολέμηση των ανισοτήτων ω μοχλός για την τόνωση της δημιουργία θέσεων εργασία και ανάπτυξης Μαρίσα Ματίας, είσαι εισηγήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Διότι μιλούμε για μια γνωμοδότηση και γνωρίζουμε όλοι ότι ε, είναι περιορισμένες ε, οι δυνατότητες ε, να επεκταθούμε. Μιλούμε για ενίσχυση της απασχόλησης, αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Απασχόλησης και όπως είπα η έκθεση του κειμένου μου έπρεπε να είναι σχετικά μικρή. Γι' αυτό και θέλω να επικεντρωθώ σε ένα θέμα που έχει σημασία από τη σκοπιά της δικής μας Επιτροπής. Δημόσιες επενδύσεις, ιδιωτικές επενδύσεις. Πολύ συχνά πρόκειται για ένα κοινωνικό ε, πρόβλημα, το πρόβλημα της ε, ανισότητας. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι πολλές φορές αυτό το φαινόμενο έχει και οικονομικές επιπτώσεις. Γι' αυτό και απαιτούνται ιδιωτικέ και δημόσιε επενδύσει, διότι μέσω των επενδύσεων δημιουργούνται θέσει απασχόληση. Ε, και η ανεργία είναι μία από τις βασικότερες πηγές ανισοτήτων. Μπορούμε να ε, ορίσουμε ε, ελάχιστες, ε, ελάχιστα όρια ε, για, την, ε, ε, για τη διαβίωση. Πρέπει να κλείσουν ε, αυτά τα, τα κενά που προκαλούν τις ανισότητες. Αν θέλουμε ειλικρινά λοιπόν να καταπολεμήσουμε τις κοινωνικές ανισότητες, ανισότητες πρέπει να έχουμε καθαρό ότι πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση είναι μια πρόκληση, αλλά είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για να γίνουν επενδύσεις. Προσπάθησα λοιπόν στην γνωμοδότησή μου να επικεντρωθώ σε αυτά τα δύο θέματα που θεωρώ ότι είναι κεντρική σημασία και φυσικά ε, ε, προσβλέπω και στην ε, συζήτηση με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Οι σκιώδεις έχουν τώρα τον λόγο. Κύριος Μπάλτς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα τοποθετηθώ σύντομα. Μια και δεν είναι εδώ και ο δισηγητής ο κ. μαντουσελο μια μια-δυο σκέψεις μου εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα σας πω. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρή Σωματεία, την συγγετριά μας, για τη δουλειά της. Με σύντομο και σαφή τρόπο και είναι θετικό αυτό. Αρκετές φορές ε, διατυπώνω τις θέσεις της μέσα σε μια πρόταση. Διαβάζω στην πρόταση αυτή. Εμένα με παρακίνησε να μελέτησω ιδιαίτερα στο ζήτημα του τι είδους ε, ανισότητες είναι αυτές στις οποίες αναφερόμαστε. Είδαμε τους τελευταίους μήνες ότι αναπτύσσεται ένας ευρύτερος διάλογος στο θέμα της ανισότητας και για μένα αυτός ο διάλογος διονκώνεται διαρκώς και μας υποχρεώνει εν τέλει να θέσουμε το ερώτημα πώς μετράμε την ανισότητα. Με ποια κριτήρια. Και κάτι άλλο σχετικό με την ανεργία ως κύριο προβλήματος. Βεβαίως η ανεργία είναι πάντα ένα σημαντικό πρόβλημα αλλά και σε αυτό το δημόσιο διάλογο και εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε ποιοι είναι οι όροι δημιουργίας θέσεως εργασίας, με ποιο τρόπο θα, τους, θα τις ενισχύσουμε. Στην ε, Γερμανία λέμε πολύ ωραία ότι κοινωνικό μέτρο είναι αυτό το οποίο γεννά θέσει εργασία. Ίσως αυτό μπορώ να συνεισφέρω εγώ στη συζήτηση, ευχαριστώντας τη Μαρία Μαρίζα Ματίας για την πρότασή της και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις προτάσεις αυτές. Είναι σημαντικό το θέμα και γι' αυτό θέλησα και να λάβω το λόγο εν συντομία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άιβαν ε, ήταν εκ μέρους των S&D στο κατάλογό μου, αλλά δεν είναι εδώ. Κύριε Τρεμόσα, ούτε εσείς είστε εδώ, αλλά ο κύριος Όζοκ είναι. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ κύριε Ματίας για το κείμενο που μας προτείνατε. Θα πρέπει να υπενθυμίσω πάντως ότι η ομάδα μας, η CR, έχει σημαντικές επιφυλάξεις σε σχέση με την έκθεση αυτή. Βεβαίως είναι σωστή η διάγνωση στην οποία προβαίνεται, δηλαδή ε, το ότι υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές δυσκολίες στις κοινωνίες μας, δυσκολία για τους νέους να εξεύρουν μια θέση εργασίας, τοξικές μορφές απασχόλησης στα όρια της νομιμότητας. Αυτά τα συμβόλαια σκουπίδια, σκύβαλα, όλες αυτές οι διαφορετικές μορφές εργασίας. Και βέβαια ρόλο των σωματείων των συνδικαλιστικών για την πραγωγή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Όλα αυτά πολύ καλά τα λέτε. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά, όσο σωστή και αν είναι η διάγνωση για το κομμάτι στο οποίο κάνετε τις προτάσεις σας για λύση, ουσιαστικά μας προτείνεται μόνο την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πέραν ε, κάθε ορίου κοινωνικής πολιτικής, με την νέα οδηγία για την αδιαμετρότητα, με τα συστήματα για την ασφάλιση ενεργείας στην Ευρώπη, με την οδηγία για τις συνθήκες εργασίας. Έχουμε εργαλεία τα οποία μπορεί να φαίνονται πολύ σωστά και απαραίτητα, ε, σε μια πρώτη ματιά, αλλά αν τα κοιτάξει κανείς πιο προσεκτικά, μάλλον θα αμφέβαλε για τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητά τους. Θα ήταν τέτοια εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ίδιο αποτελεσματικά με ε, το επίπεδο που θα μπορούσαν να προσφέρουν σε εθνικό επίπεδο. Δεν νομίζω, γιατί σε εθνικό επίπεδο γνωρίζει κανείς πώς είναι η αγορά και πώς περιγράφονται αλλά και περιορίζονται τα προβλήματα. Πολύ συγκεκριμένα μπορεί να δώσω κάποιες προτάσεις από την πολωνική κυβέρνηση, η οποία έχει προβεί σε ένα ευρύτατο πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης των οικογενειακών με ένα μόνο παιδί και που μάλιστα υιοθέτησε, ε, ε, υιοθέτησε μέτρα που βελτίωσαν σημαντικά την κατάσταση των ε, οικογενειών που είχαν δυσκολίες και μάλιστα υποστήριξε και βοήθησε και οικογένειε που βρίσκονται στον κίνδυνο τη περιθωριοποίηση. Δεν νομίζω όμω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν αντίστοιχα μέτρα να φέρουν αποτέλεσμα. Άλλωστε και η Διασηγήτρια παραδέχεται πω το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν έχει διαδραματίσει το ρόλο που αναμενόταν ότι θα διαδραματίσει ω προ την επανεξισορρόπηση των ευκαιριών, των ίσων ευκαιριών. Δηλαδή δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τότε γιατί να προάγουμε περισσότερη εναρμόνιση, γιατί να προτείνουμε περισσότερα μέτρα εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όλα αυτά χωρίς να συζητούμε τα αποτελέσματα των πιλωτικών προγραμμάτων. Ελπίζω ότι θα ληφθεί υπόψη η ε, επιφυλακτικότητα αυτή της ομάδας μου, γιατί θα την καταγράψουμε στις θέσεις μας για τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ κύριο Ζωρόκ, δεν βλέπω ε, από, την, από κανέναν. Εκ μέρους των Πρασίνων ο κύριος Γκίγκολτ, Ζέν. Μεταφέρω τους χαιρετισμού στους σκιώδου μας, στους σκιώδους μας, κυρίου Λάμπερτς. Και σημειώνω πως ε, χαιρόμαστε για τη γνωμοδότηση αυτή. Στη γνωμοδότηση, και το υπογραμμίζω, υπογραμμ... ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία θέσεων εργασία. Όσο και αν δεν συμφωνώ πως ε, οτιδήποτε παράγει η θέση εργασίας είναι μέτρο κοινωνικό, γιατί και η δουλεία θα μπορούσε έτσι να υπαχθεί στον ορισμό της ε, κοινωνικής δραστηριότητας για την παραγωγή θέσεων εργασίας για το συνάδελφο Μπάλτς και, τη γερμανική, και τον περιγερμανισμικό ορισμό του τι σημαίνουν κοινωνικά μέτρα. Α περιοριστούμε όμω στι δικέ μα εξουσίε, γιατί πολλά από τα θέματα που εγείρονται στη γνωμοδότηση δεν έχει αρμοδιότητα η Επιτροπή μα. Ε, αν διερωτηθούμε λοιπόν πού έχουμε αρμοδιότητες, πού έχουμε εξουσίες με την έκθεση της ΕΜΠΛ ή ενόψε της έκθεσης της ΕΜΠΛ, θα έλεγα καταρχάς καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και άρα απελευθέρωση των δημοσίων επενδύσεων και διευκόλυνση ορθολογικών δαπανών, ταυτόχρονα συμβάλλοντας στον περιορισμό των ανισοτήτων. Δεύτερον, ε, αν είναι πάρα πολύ άνηση η κατανομή του πλούτου με, πάρα πολλού, με κάποιους πλούσιους που έχουν πολύ χρήμα να ρίξουν στη χρηματο οικονομική αγορά, χρηματοπιστωτική αγορά και έτσι μπορούν να συμβάλλουν με τη συμπεριφορά τους στην χρηματοπιστωτική αστάθεια και άρα εδώ έχουμε ακόμη ένα παράγοντα ανισότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα συγκεκριμένα και επίσης αρμοδιότητα που έχουμε στην, στην πολιτική του ανταγωνισμού η οποία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για, τον, ε, για τη συγκράτηση των τιμών και την ε, καλύτερη απόδοση της επένδυσης του χρήματος που δαπανά κανείς, άρα προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή. Άρα θα ήταν χρήσιμες τροπολογίες οι οποίες θα συνέδεαν περισσότερο τη γνωμοδότηση με, τον, με τους τομείς αρμοδιότητων της δικής μας Επιτροπής. Ευχαριστώ Σβέν, δεν ζητεί κανείς άλλο το λόγο. Η εισηγήτρια για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω άλλη μια φορά και να τα πω κάπως τηλεγραφικά. Σε αυτά που είπε ο Μπούρκαρτ, για, τον, για το είδος ε, της ανισότητας την οποία συζητούμε, μα το είπα εισηγητικά. Όταν κανείς ε, συντάσσει μια γνωμοδότηση και όποιος έχει συντάξει γνωμοδότηση το ξέρει, ε, ε, οφείλει να ε, αυτοπεριορίζεται ως προς την έκταση του κειμένου. Εγώ προσπάθησα λοιπόν να επικεντρωθώ ε, στις ανισότητες, στην απασχόληση και στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Φυσικά και δεν αρκούν αυτά. Είναι δεδομένο αυτό. Για αυτά που είπε ο συνάδελφος από το ECR. Μα δεν είναι δική μου ε, έκθεση ο Χάβι Από την Επιτροπή Απασχόλησης είναι εκείνο που ε, θα συντάξει την έκθεση. Και εκεί εκείνος δεν κάνει καν ε, αναφορά στε, στην, στις άδειες μητρότητας σε εκείνον να τα απευθύνετε αυτά που είπατε. Εγώ απλώς μια γνωμοδότηση ε, συντάσω. Ε, αυτό δεν ήταν δικό μου σφάλμα. Ο Χάβι ε, τα, τα, έχει γράψει αυτά. Ως προς αυτά που είπε ο Σβέν, προσυπογράφω απόλυτα. Αλλά όπως είπα και νωρίτερα, σε ένα θέμα μπορούσα να, να επικεντρωθώ. Οι επενδύσεις είναι ένα θέμα που με απασχολούν πολύ. Φυσικά ε, είναι σημαντικά θέματα η φοροαποφυγή, η φορολογική απάτη, η φοροδιαφυγή, η δίκαιη κατανομή του πλούτου και του εισοδήματο. Όλα αυτά είναι σημαντικότατα θέματα, αλλά όπως καταλαβαίνετε είχα ήδη ε, υπερκαλύψει το, την έκταση του κειμένου μου. Αν θέλετε βέβαια με τροπολογίες όλα αυτά μπορούν να διορθωθούν. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα να σας πω ότι, ότι η βοηθός μου ε, εγκαταλείπει το, το γραφείο μου ε, η οποία με έχει βοηθήσει από το 2009 πάρα πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τη Ριάννα ε, το ίδιο και ολόκληρη η Επιτροπή. Ε, Οικονομικών και Νομισματικών Επιθέσεων. Και όπως είπα, πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνω πλέον. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Λάμπερτς μου έχει το λόγο, πρόεδρε. Λυσμόνισα την κάρτα μου. Είναι καθοδόν, αλλά δεν θα την έχω έτοιμη. Ευτυχώς που δεν την έχεις δέσει γύρω από το λαιμό σου, λέει ο πρόεδρος, γιατί αλλιώ δεν μπορούσε να την αφήσει πουθενά. Έτσι μου λέει ο δασκαλό μου όταν έχανα τη γόμα στο σχολείο. Και έχουμε να ανατρέψουμε τη σειρά, γιατί ο συνάδελφος θα πρέπει να φύγει, δεν έχετε αντιρρήσεις. Έχετε όλοι τις κάρτες σας, βιέγκας. cum tempore, όπως λέμε στα λατινικά. Δοκιμαστικά. Πλην του κύριου Λάμπερτς, έχετε όλη την κάρτα σας. Ας αρχίσουμε λοιπόν δοκιμαστική ψηφοφορία. Α, εντάξει, εδώ είναι. Ωραία, είναι ανοιχτή η ψηφοφορία λοιπόν, δοκιμαστική. Οι πράσινοι δεν έχουν ε, παραπάνω ψήφους από ό,τι πρέπει να μετρήσουμε. Εντάξει, καλά πάμε στη δοκιμή. Πέρας λοιπόν της δοκιμαστικής, με το σχέδιο γνωμοδότησης για τις ελάχιστες πολιτικές, για τις πολιτικές περιαλλαχές του εισοδήματος του εργαλείου για την κατοικολόμηση της φτώχειας, Εμβαστική H, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται Τροπολογία 74 υπέρ. Κατά. Ας το επαληθεύσουμε. 74, τέσσερα, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία, πέρας. Και εγκρίνεται. 75 υπέρ. 23 υπέρ, 21 κατά. Ε, ό,τι μου λέει οθόνη κάνω, δεν ε, έχω πρόσβαση στην ε, υψηλή τεχνολογία. Να το βγάλεις κλωδία και την άλλη φορά στην οθόνη. 75 λοιπόν υπέρ κατά αποχές με την ίδια πλειοψηφία 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ ε, του Υπουργού που παρετήθη υπέρ αποχές και της Υπουργού που παρετήθη. Ναι, το διάβασα στις ε, γαλλικές εφημερίδες. Πάντως, Πρόεδρε, δεν ήταν ούτε αστείο, ούτε και σωστό αυτό που κάνατε. Καλά, 78 υπέρ κατά. Ας το επαληθεύσουμε. 78 υπέρ Μάλλον ανοίγει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική γιώτα, αι, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές. Απερίφθη. 91 υπέρ, κατά. Το επαληθεύουμε ή τελώσουν οι πλειοψηφίες. Άρχεται η αλλάζουν Με μία ψήφο διαφορά. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Να επαληθεύσουμε. 93. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Εντάξει. Μικρή υπερψηφία, αλλά ορατή. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές με την ίδια πλειοψηφία. Εγκρίνεται 95 υπέρ. Κατά Αποχές σας επαληθεύσουμε τώρα. 95. Ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ε, J υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 108. Απορρίπτεται. Αποχές και επαληθεύουμε την 108. 108 λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται συμβιβαστική και η κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 121 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 122 υπέρ κατά αποχές οι σοσιαλιστές τι κάνουν καλά ε, ηλεκτρονικά 122 αρχής ψηφοφορία ναι, τώρα είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ναι. Πέρας και έγκρινεται. 124 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη 125 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική L λάμδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. M μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απερίφθη, ας το δούμε όμως, 143 ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ναι, καλά έκανα και το έλεγξα. Απερίφθη όμως. 145 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 146 υπέρ κατά αποχές μάλλον έχει εγκριθεί αλλά ας την επαληθεύσουμε 146 αρχής ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 148 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 149 έχει αποσυρθεί. 150 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται 140, 152 υπέρ, κατά. Α, Α την απολυθεύσουμε και νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Αρχίζει η ψηφοφορία 152. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές απεριφθεί. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική νη 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 6 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη. 22 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 23 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε 23 ψηφίζουμε η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας και απερίφθη αυτό δεν μπορούσα να το δω 24 34 υπέρ κατά αποχές ναι εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ. Ναι, ναι, εγκρίθηκε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 34 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 43 υπέρ. Κατά. Για να επαληθεύσουμε την 43 παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 44 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 45 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 47 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 48 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 49 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 50 υπέρ κατά αποχές για να το επαληθεύσουμε. Την 50 παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 56 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ας επαληθεύσουμε τη 57 λοιπόν. Και αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές με την ίδια πλειοψηφία και εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε την 60 αρχίζει η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι Πέρας. Απερίφθη. ψηφία, Συμβαστική F υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και φτάνω στην τελική ψηφοφορία έτσι. Ονομαστικά. Ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν η τελική. Αρχίζει. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τώρα ελπίζω να προλάβεις και την σου. Και τώρα γυρνούμε πίσω στο προηγούμενο θέμα. Σχέδιο γνωμοδότησης προς ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο καλυμμένων ομολόγων με τον κύριο Λούκε. Συμβαστική πρώτη. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Σ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι η 63 απεσήρθη ήταν δική σου. Ωραία. Άρα περνάμε στην 74 ως προσθήκη στην συμβαστική D. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα μπορώ να περάσω στην συμβαστική E, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική F, προσεκτικά. Ο πρόεδρος, όχι εγώ, είπε ότι πρέπει πρώτα να ψηφίσουμε επί του FBs. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο πρόεδρος πρέπει πάντα να έχει δίκιο, αλλά τέλος πάντων. FBs, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρα δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε επί της F. Συμβαστική G, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στις ιδεολογικές σκέψεις υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Recital. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία για την τροπολογία 5. Υπέρ σοσιαλιστές το ζήτησαν. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ωραίο αυτό. Και πάμε στην τελική ψηφοφορία, ονομαστικά, όπως πάντοτε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά για το σύνολο της ε, έκθεσης του κυρίου Λούκε, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 43 υπέρ, Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά για το έργο σας και ελπίζουμε η Κομισιόν να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της μετά την υιοθέτηση της και στην Ολομέλεια. Επόμενο θέμα. Τέλος των ψηφοφοριών. Έλεγχος κατεξοδότηση πράξεων και εκτελεστικών μέτρων. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μέτρα IFL επίπεδο 2 για τον κανονισμό για τις διατραπεζικές προμήθειες. Ο εισηγητής μας, ο Παύλο, μας έχει εγκαταλείψει, γι' αυτό και εγώ έχω την τιμή να τον εκπροσωπήσω. Βρισκόμαστε πλέον στην 31η εβδομάδα για, την, για τον έλεγχο των κεστοδότησης πράξεων και των εκτελεστικών μέτρων. Σήμερα θα συζητήσουμε για ε, τα, ζητήματα που σχετίζονται με το ε, πρότυπο, το διεθνές πρότυπο για τις πληρωμές με κάρτα και τις, ε, τους φορείς επεξεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή εξέδωσε το πρότυπό της Πέρση, τον Ιούλιο στις 5 Ιανουαρίου 2017 προτείναμε 5, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πέντε τροποποιήσεις στο κείμενο της EBA ε, με στόχο την ενίσχυση της απέτησης ανεξαρτησίας. Η EBA συμφώνησε με τρεις από αυτές τις αλλαγές, αλλά διαφώνησε με τρεις επίσης καθώς το ΆΕΦΑΡ δεν απαιτεί νομικό διαχωρισμό των ε, φορέων. Πρώτο θέμα που μας απασχολεί είναι ο διαχωρισμός, ο, ο, η συμμετοχή των εργαζομένων συμμετοχές ε, και η επενδυματική πολιτική και τρίτον οι προϋποθέσεις για τις διευθυντικές σχέσεις που καλύπτονται από το ίδιο άτομο σε ένα διοικητικό όργανο. Είναι ενημέρωση, σας, έχουμε ενημερώσει και γραπτός μέσω της γραμματείας. Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Μαρία Βαλέντσα από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και τον Ντίλ Κάουμπριχ από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή που είναι τμήματάρχης για την, για την προστασία των καταναλωτών και την καινοτομία και θέλω να σας δώσω το λόγο για να μας κάνουν μια σύντομη παρουσίαση. Πέντε λεπτά συνήθως δίνουμε και από εκεί και πέρα θα έχουμε έναν κύκλο ε, με τοποθετήσεις από τους εισηγητές, κοιόδης εισηγητές και ερωταπαντήσεις. Ξεκινώ με την Κομισιόν, αν δεν έχετε αντίρρηση. Οπότε, κύριε Βιλάντσα, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, πολύ. Δεν θα μπω σε πάρα πολλέ λεπτομέρειες. Είναι ένα θέμα το οποίο έχετε δει γιατί έχουμε μοιράσει το σχετικό σημείωμα. Έχουμε για την ανεξαρτησία της αλλαγής που έχουμε στην νομοθεσία και το μέτρο αυτό έχει ως σκοπό να αλλάξει τις ε, κάθετες πληρωμές στους φορείς διεκπαιρέωσης πληρωμών για τις πιστωτικές κάρτες. Και ο στόχος ε, αυτού του πρότυπου που είναι κανονιστικό και ρυθμιστικό είναι να καλύψουμε αυτές τις καθετοποιημένες ε, περιπτώσεις Αν μιλάμε για τη διάκριση των διαφόρων ε, ε, ε, πιστοτικών από τους φορείς που διεκπεραιώνουν τις πληρωμές, ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι περισσότερες από αυτές τις οντότητες, που νομίζω ότι είναι 28 από τις 31, ήδη έχουν εφαρμόσει αυτή τη διάκριση. Οπότε αυτό που προτείνουμε εδώ είναι μια ποσοτικοποίηση των όσων συμβαίνουν σήμερα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κλάδου. Αντίθετα, οι διεθνεί παίκτε όπω η Visa και η Mastercard αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζουν αυτή τη διάκριση, τουλάχιστον όχι ακόμα, οπότε η πρότασή μα ουσιαστικά έχει ε, στόχο να ξεπεραστούν κάποιες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό από διεθνείς παίκτες που δρούν στην, ε, και επιχειρούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Και με αυτά κατά νου, θα μπω και στα πιο συγκεκριμένα για αυτές τις τρεις τροπολογίες όπου έχουμε διαφορές με την ΙΜΠΑ. Μην ξεχνάτε πως η συνεργασία μαζί τους είναι εξαιρετική, οπότε είναι μικρά τα σημεία στα οποία έχουμε απόκληση απόψεων, γενικότερα πάντως για τις βασικές αρχές συμφωνούμε. Κοινούς παρανομαστής για τα τρία σημεία που μας ανησυχούν. δίνουν παρεκκλήσεις οι οποίες δεν προβλέπονται στον κανονισμό επίπεδου 1. Στον κανονισμό εκεί το κείμενο είναι ξεκάθαρο. Η απέτηση υπάρχει για την ανεξαρτησία των λογιστικών αποφάσεων και δεν προβλέπεται οποιαδήποτε παρέκκληση. Η έχει βρει στήριξη για την πρόταση αυτή για παρέκκληση από άλλες ε, ε, σχετικές ε, χρηματοπιστωτικές οδηγίες, αντιμήφετ, όπου η παρέκκληση επιτρέπεται και για το πρώτο επίπεδο, όχι μόνο για το επίπεδο 2. Οπότε εδώ νομίζω ότι εσείς ως συνομοθέτης θα πρέπει να διατηρήσετε τα προνομιά σας και να το αφήσουμε ως έχει. Τώρα, για τα τρία σημεία που μας ανησυχούν. Καταρχήν, άρθρο 13 η προτινόμενη παρέκκληση για την ανεξαρτησία του προσωπικού σε περίπτωση νέων εκαθαρίσεων. Εδώ προτείνουν μια παρέκκληση έτσι ώστε να προβλέπετε αυτή η παρέκκληση από την ανεξαρτησία σε περίπτωση καινοτομίας και ακολουθούν το εξής σκεπτικό. Δηλαδή, αν δεν επιτρέψουμε στο προσωπικό να εξαιρεθεί λόγω καινοτομία, μπορεί τελικά για τις μεγαλύτερε οντότητες να αποτελεί ένα, μια δια, ε, στρέβλωση. Αυτό βέβαια ευνοεί τις καθετοποιημένες οντότητες σε σχέση με τους ανεξάρτητους ε, διεκπαιρώτες που άρα ευνοεί ουσιαστικά εταιρείε όπως η Visa και η Mastercard οι οποίες είναι έτσι καθετοποιημένες. Οπότε δεν θέλουμε αυτή την παρέκκληση γιατί έτσι κι αλλιώς ε, για το πρώτο επίπεδο δεν επιτρέπεται. Τώρα, για το διεθνή ανταγωνισμό να σας πω πως δεν πιστεύουμε πως υπάρχουν άλλοι παίκτες στον κόσμο που θα επιτρέψουν τέτοιου είδους καινοτομίες. Τουλάχιστον όχι προκρίνοντας τέτοιου είδους ε, παρεκκλήσεις χάρη καινοτομία, γιατί όλοι οι παίκτες, είτε είναι ευρωπαϊκές εταιρείε είτε θεατρικές στην ευρωπαϊκή επικράτεια, θα πρέπει να εφαρμόσουν τους ίδιους κανόνες. Οπότε αυτό που θέλουμε να καλύψουμε εδώ είναι οι μεγάλοι διεθνείς παίκτες, Visa, Mastercard κτλ. Για το δεύτερο θέμα, άρθρο 11.3, δηλαδή συμμετοχή προσωπικού σε όλα ε, τα μπόνους, ε, τα κατοχή μετοχών κτλ. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Αυτό συμμορφώνεται με το πρώτο επίπεδο. Γιατί εδώ μιλάμε για πλήρη ανεξαρτησία χωρίς καμία παρέκκληση στο επίπεδο αυτό και θεωρούμε πως αν εισάγουμε εδώ μια παρέκκληση, η προτινόμενη παρέκκληση θα δημιουργήσει κίνητρα για το προσωπικό τα οποία ε, εργάζονται σε ένα κομμάτι της επιχείρησης να ε, ε, κάνουν διακριτική μεταχείριση οικονομική για το υπόλοιπο. Αυτή η λειτουργική διάκριση έχει λειτουργήσει σε άλλους κλάδους, στις τηλεπικοινωνίες, στην ηλεκτρική ενέργεια, όπου είπαμε πως η δημιουργία αυτών των σχεδίων συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των εργαζομένων είναι εύκολη, δεν είναι εξαιρετικά περίπλοκη για τις εταιρείες, οπότε εκεί έχει επιτραπεί. Η προτινόμενη παρέκκληση έρχεται σε αντίφαση με την απαγόρευση που υπάρχει που είναι τα άρθρα 11.1 και 11.2 του κανονιστικού ε, κανονισμού για τα τεχνικά πρότυπα, όπου υπάρχει σχετική διάταξη που δεν επιτρέπει άμεση ή έμεση ε, σχέση με την αμοιβή του άλλου τμήματος της νομικής οντότητας. Οπότε η πρόταση αυτή για παρέκκληση θα δημιουργούσε μία αντίφαση με το ίδιο το κείμενο. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, 16.1 ανεξαρτησία των διαχειριστικών ε, φορέων και ο αριθμός ε, διευθυντικών στελεχών. Νομίζω πως εδώ χρειάζεται μια, ένας ποσοτικός ε, περιορισμός, αλλά αυτός που έχει τοποθετηθεί εδώ αυθαίρετα δεν μας ικανοποιεί. Χρειάζεται να πάνε κάποια αντιμηνικά κριτήρια που να ορίζουν τον αριθμό αυτό. Και τέλος για την ε, λειτουργική ε, σε αντιδιαστολή με την επιχειρησιακή διάκριση σε όλες τις διατάξεις εμείς μιλάμε για λειτουργική διάκριση αυτή είναι η συμφωνία στο επίπεδο 1 δεν μίλησαμε ποτέ για νόμιμη, νομική ε, διάκριση που σημαίνει δημιουργία διαφορετικών οντοτήτων ποτέ δεν το ζητήσαμε εμείς μιλάμε για διάκριση μεταξύ επιχειρηματικών επιχειρησιακών μονάδων, οικονομική διάκριση, διάκριση στρατηγικής κτλ. Αλλά ποτέ δεν ζητήσαμε να υπάρχει νομική διάκριση μεταξύ αυτών. Οπότε το λέω τώρα και θέλω να το λάβετε δεόντως υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος του κύριο Χάμπρικ από την EBA. Ευχαριστώ. Ξέρετε πρόεδρε, από τα μέλη της Επιτροπής σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να σας εξηγήσουμε είναι το δικό μα σκεπτικό. Πρώτον, να συμφωνήσω με αυτά που είπε η συνάδελφος από την Κομισιόν. Έχουμε τρία ζητήματα ε, ε, τα οποία, ε, στα οποία η, η άποψή μας είναι διαφορετική από τις Κομισιόν, ωστόσο μέσω τη συνεργασία μας έχουμε προχωρήσει τους τελευταίους μήνες. Ας δούμε λοιπόν αυτές τις τρεις τροπολογίε που πρότεινε η Κομισιόν και με τι οποίε εμεί διαφωνούμε. Και πάλι, να ξεκινήσω με την πρόταση της Κομισιόν τα συστήματα πληρωμής με κάρτας και, το, και τους φορείς επεξεργασίας να μην ε, ταυτίζονται προκειμένου να μην υπάρχει αθέμητο ε, πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό ε, δεδομένου ότι τα συστήματα πληρωμής με κάρτας έχουν πρόσβαση σε ε, πολλές δυνατότητες. Ε, ε, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και διεθνείς φορείς οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν και πόρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δεν ισχύει ο κανονισμός. Αυτή είναι η άποψη της EBA να επανεισαχθεί αυτή η παράγραφος που διαγράφει από την Κομισιόν ωστόσο συμφωνούμε με την ανησυχία της Επιτροπής και γι' αυτό τον λόγο εμείς προτείνουμε να αποσαφηνίσουμε την ε, σύνδεση με τις απαιτήσει που σχετίζονται με τα άρθρα 11 και ιδίως την ε, υποχρέωση να μην αποκαλύπτονται επιστευτικές προφορίες. Όσον αφορά την τροπολογία που σχετίζεται με τα, με τις, ε, με τα γενικά επιδόματα, την επιδοματική πολιτική, το άρθρο 11 του RTS, η Κομισιόν θεωρεί ότι αυτό είναι ε, ε, ασύμβατο με τα συστήματα αποδοχών, δεδομένου ότι οι αποδοχές ε, των εργαζομένων μπορεί να εξαρτώνται από τις επιδόσεις του φορέα επεξεργασίας, για τον οποίο όμως εκείνος δεν εργάζεται, οι εκείνοι οι εργαζόμενοι δηλαδή δεν εργάζονται. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι Συγγνώμη να βρω λίγο τη σελίδα μου. Just, στην επόμενη τροπολογία και θα σας τα πω μετά. Ε, που είναι η πρόταση Κομισιόν να αναδιατοπαθούν τα σαφή και αντικειμενικά κριτήρια. Εδώ διαφορούμε με την Κομισιόν, διότι το RTS συμπεριλαμβάνει ήδη σαφή κριτήρια και απαιτήσει και γι' αυτό και αποκαταστήσαμε αυτή την παράγραφο που προτάθηκε να διαγραφεί από την Κομισιόν. Όσον αφορά την άποψη που εξέφρασε μόλις η Κομισιόν σχετικά με το RTS μας και ότι ε, δημιουργεί μια εξαίρεση στο κείμενο του επίπεδου 1, εμείς διαφωνούμε με αυτή την άποψη. Θέλουμε να εξασφαλιστεί ότι είμαστε εντός του πλαισίου που ορίζει ο νόμος, γιατί εμείς δεν είμαστε νομοθέτες και η απόκληση για, ε, όσον αφορά την ανεξαρτησία ε, θα υπήρχε αν ε, οριζόταν η ανεξαρτησία στην, στην νομοθεσία επίπεδου 1. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Το RTS καλείται να ορίσει τι ακριβώς είναι η ανεξαρτησία. Γι' αυτό και δεν θεωρούμε ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με κάποιο είδους εξαίρεσης. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ να περάσουμε στον εισηγητή. Θα μιλήσω γερμανικά. Θέλω να ασχοληθούμε σήμερα με τρία θέματα. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Όσον αφορά την ανεξαρτησία του προσωπικού στον τομέα της έρευνας και της κοινοτομία, εδώ η EBA ε, προτείνει τον αυστηρό ε, όσον αφορά τον αυστηρό διαχωρισμό να επιτρέπεται μια εξαίρεση για την έρευνα και την καινοτομία. Γιατί αυτό θα δώσει τη δυνατότητα κατά τη γνώμη της στις μικρές επιχειρήσεις να ε, προχωρήσουν στο έργο τους, ε, στην έρευνα και στην καινοτομία. Όσο μεγαλύτερη μια επιχείρηση, όσο περισσότερους εργαζόμενους μπορεί να διαθέσει στην έρευνα, τόσο καλύτερα είναι και τόσο καλύτερες είναι και οι επιδόσεις της. Γι' αυτό ε, και η αγορά που σήμερα κυριαρχείται ε, από μεγάλες εταιρείες ε, που μπορούν φυσικά να ανταποκριθούν σε, μια τέτοια, ένα τέτοιο διαχωρισμό και να δραστηριοποιηθούν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. η κατάσταση είναι αυτή. Αν θέλουμε όμως μεγαλύτερες και περισσότερες καινοτομίες στον τομέα των πληρωμών, και αυτό ήταν και η δική μας πρόθεση, χρειαζόμαστε ευνοϊκές διατάξεις ε, όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις και στο, στο, στο θέμα αυτού του αυστηρού διαχωρισμού. Ερώτημα λοιπόν προς τον Κομισιόν. Πώς μπορούν να εξελιχθούν οι πληρωμές με κάρτα και εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν, αν δεν θεσπίσουμε εμείς ένα ε, ευνοϊκό καθεστώς όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων στις μετοχές ε, και τις, ε, υποχ... τις... Ε, ορίζεται από την EBA να υπάρχει εξαίρεση για αυτές τις εταιρείες. Η Κομισιόν απέριψε όμως αυτή την πρόταση της EBA. Ωστόσο στο επίπεδο 1 δεν μιλούμε για κατάτμιση των επιχειρήσεων, αλλά για οργανωτικό διαχωρισμό. Ιδίω για τι μικρέ επιχειρήσει θα ήταν δυσανάλογο για κάθε τμήμα τη επιχείρηση να υπάρχει ε, ξεχωριστό πρόγραμμα ε, συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο των εργαζομένων. Πώ θα μπορούσαν να ξεπεριστούν αυτά τα εμπόδια, λοιπόν, πώ θα μπορούσαν να δοθούν αυτέ τι δυνατότητε και στι μικρέ επιχειρήσει χωρί να επιβαρύνονται με αυτό το διοικητικό άχθο. Και τέλο, όσον αφορά τις διοικητικές θέσεις που μπορούν να καλύπτονται, αν μπορούν να καλύπτονται από το ίδιο άτομο. Η πρόταση ε, της ΕΜΠΑ είναι να υπάρχει διαχωρισμός ε, και να υπάρχει ανώτατο όριο των, ε, του αριθμού των διοικητικών θέσεων που μπορεί να καλύπτονται από το ίδιο άτομο. Εδώ έχω τις αμφιβολίες μου ως προς την πρόταση αυτή η αιτιολογική σκέψη 33 αναφέρει ότι τα συστήματα πληρωμής με κάρτα και οι οντότητες επεξεργασίας θα πρέπει ανεξάρτητα μεταξύ τους να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους και αυτό ε, δεν εξυπηρετείται απλά και μόνο με ένα αριθμητικό, όριο των ε, διοικητικών ε, θέσεων που μπορεί να καλύπτει κανείς. Θεωρεί η EBA ότι είναι επαρκής λοιπόν η πρόταση της. Ε, η Κομισιόν πρότεινε να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος δύο ετών προκειμένου να καθοριστούν οι διευθυντικές θέσεις και πώς θα στελεχωθούν αυτές. Είναι πράγματι Κομισιόν ε, αυτό το χρονικό διάστημα ε, κατάλληλο και ενδεδειγμένο. Είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα αυτό και η αγορά είναι αρκετά μικρή. Δεδομένου μάλιστα και ε, του περιορισμού ως προς την ελευθερία άσκηση του επαγγέλματο, μήπως ε, Κομισιόν η πρότασή σας αυτή δεν είναι αναλογική. Αυτά και επανέρχομαι στην ιδιότητά μου ως Προέδρου, επιστρέφω στα αγγλικά να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο σοσιαλιστών, τον Όλη Λούντβικσον. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω τα εξή για την EBA. Έχουν δημοσιευθεί αυτά τα τεχνικά πρότυπα για τη διάκριση μεταξύ των οδητών διεκπαιρέωσης και των πιστοτικών ε, των εταιριών πιστοτικών καρτών και όλα αυτά τα έχουμε στο άρθρο 7.1 του σχετικού κανονισμού. Και τέτοιου είδους συστήματος πληρωμής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα από τις εταιρείες εκαθάρισης ή διεκπαιρέωσης όταν μιλάμε για την διεκπαιρέωση της πληρωμής τουλάχιστον ε, σε επίπεδο λογιστικής. Στον ίδιο τον κανονισμό εξασφαλίζουμε πως αυτό γίνεται διακριτά έτσι ώστε να προωθήσουμε την καινοτομία όμως, στην πρόταση αυτή δεν βρίσκουμε καμία στήριξη από τον ίδιο τον κανονισμό είτε στα εκτιμώντας είτε στο 7. Δηλαδή, θα πρέπει αυτά τα δύο να διακρίνονται μεταξύ τους όταν κάνει κανείς κάποιες αποφάσεις, όταν παίρνει κανείς αποφάσεις στο, σε οργανωτικά ή σε λογιστικά θέματα. Μην ξεπερνάμε την ίδια μας την εντολή. Αυτές οι παρεκκλήσεις δεν πρόκειται να διευκολύνουν τους νέους παίκτες να μπουν στην αγορά ούτε πρόκειται να τους βοηθήσουν στο να εμφανιστεί περισσότερος ανταγωνισμός. Όχι. Μόνο οι καθετοποιημένες ε, μονάδες, οι καθετοποιημένες εταιρείε, που είναι οι πολύ μεγάλες θα ευνοηθούν, γιατί έτσι κι, αλλιώς, έτσι κι αλλιώς αυτές κυριαρχούν στην αγορά. Οπότε νέους παίκτες δεν θα δούμε. Και προτάθηκε και μία παρέκκληση για το προσωπικό το οποίο εργάζεται έτσι ώστε να υπάρχει ένα είδος λειτουργικής ε, διάκρισης. Όμως, ο κανονισμός νομίζω το λέει απερίφραστα, γιατί έχουμε το εκτιμώντας 33, το οποίο λέει πως δεν μπορεί να έχουμε ε, αυτά τα κοινά ε, προγράμματα bonus, θα πρέπει να υπάρχει μια διακριτή οργάνωση και αυτό τονίζεται και πάλι στο 7 άρα λοιπόν δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παρέκκληση αυτή δεν ευθυγραμμίζεται και δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσει που υπάρχουν για οργανωτική ανεξαρτησία και αυτονομία. Δηλαδή το 16.1. Δηλαδή η πρόταση της EBA ε, δεν συμμορφώνεται ούτε με το 11.1 ούτε με το 11.2 που έχουμε στα τεχνικά πρότυπα που απαιτούν ανεξαρτησία οργανωτική. Οπότε, ε, για τα διοικητικά συμβούλια, για παράδειγμα, για τα διευθυντικά στελέχη. Νομίζω ότι είναι ε, ε, ξεκάθαρα και έχουμε και το εκτιμώντα 43 του κανονισμού, όπου ορίζουμε πως αυτά τα είδη πληρωμών μέσω πιστοτικών καρτών και οι οντότητε διεκπαιρέωσης των πληρωμών δεν μπορούν να έχουν κοινή διαχείριση. Άρα λοιπόν η πρόταση που γίνεται δεν μπορεί να ε, συμμορφωθεί με το 16.1 για τις τεχνικές προδιαγραφές που μιλάμε για τεχνική ανεξαρτησία. Και αυτοί οι επικαλυπτόμενοι κανόνες δεν νομίζω πως εξασφαλίζουν έτσι όπως προτείνεται την ανεξαρτησία μεταξύ των δύο αυτών αντοτήτων. Θα περάσω το... Ευχαριστώ. Προσπαθώ να δω ποιος από τους συναδέλφους έχει μείνει εδώ. Δεν είναι εδώ ο κύριος Άσλι Φόξ ή άλλος από το ECR, ούτε από τους φιλελευθέρους, ούτε την κυρία Μακάρθη, από την ΚΟΕ, ούτε άλλον. Άικχαουτ από τους πράσινους ή άλλος πράσινος δεν υπάρχει. Ούτε και το Μάρκο βλέπω, η FTD, ή άλλον από το EFTD. Και άρα δεν χρειάζεται να ζητήσω. Ποιος θέλει το καρσιδιά, όλοι. Όχι, δεν κανείς πρέπει να πω ότι απογοητεύομαι, διότι στις συνεδρίες των Σκιωδών είχε στήσει να, είχαν στήσει όλοι να γίνει αυτή, αυτός ο έλεγχος. Και να είναι εδώ η Κομισιόν, όπως τους είδαμε σήμερα. Θα το εγείρω το θέμα στην προσοχή συνεδρία των Σκιωδών. Αλλά συγχαίρω τον Όλε, που είναι ο τελευταίος που στάθηκε στο ύψος. Και εγώ επειδή είμαι πρόεδρος αναγκαστικά. Αλλά πολλά ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Να ακούσουμε πρώτα την Επιτροπή και μετά την ΕΜΠΑ. Κυρία Φορέντσα. Ναι, ένα-ένα θα απαντήσω. Διεθνή συστήματα καρτών πλήρωμες, έχουν ε, ενοποιηθεί κατακόρυφα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ένα πεδίο ισότιμου ανταγωνισμό μεταξύ Ευρωπαίων ε, και φορέων που δραστηριοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο ΣΕΠΑ, αυτορυθμιζόμενη πρωτοβουλία, τα περισσότερα από τα συστήματα, 28 από τα 31 συγκεκριμένα συστήματα καρτών, πληρωμές έχουν κάνουν αυτή τη λειτουργική διάκριση, το διαχωρισμό. Άρα αυτό που κάνουμε περισσότερο είναι η κωδικοποίηση της υφιστάμενης στην ε, τωρινή κατάσταση της αγοράς της Ευρώπης ε, κατάστασης. Απαιτήσει διαχωρισμού διεθνής φορείς που ισχύει βέβαια και για τις διεθνείς, για τα διεθνή συστήματα, γιατί εφαρμόζονται όταν οι πληρωμές μάλλον ο πάροχος πληρωμών, υπηρεσιών πληρωμών του αγοραστή ή του πληρώνοντος και ο ε, πάροχος υπηρεσιών πληρωμής του ε, πληρωνομένου βρίσκονται στην Ευρώπη. Visa, Mastercard, Mastercard ή κάποια άλλη ευρωπαϊκή εταιρεία. Ε, Λειτουργική διαχωρισμός και λάφρυνση του φόρτου. Δεν έχω εντολή βέβαια να συζητήσω κάτι άλλο σήμερα μαζί σας. Αλλά στη διαδικασία που έχουμε ήδη ανοίξει βλέπουμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα προβληματικός ο διαχωρισμός των σχεδίων μετοχών των εργαζομένων. Το βλέπουμε και στις τηλεπικοινωνίες και σε άλλα στήματα. Αντίστοιχα σε κλάδους ε, που είναι ενοποιημένα αυτά τα συστήματα και δεν βλέπουμε ιδιαίτερες δυσκολίε ή διαφορές. Και άρα πιστεύουμε ότι και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε στην, ε, στον κλάδο των καρτών πληρωμών που είναι καινούριο σχετικά. Ο διαχωρισμός πάντως διαφόρων δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Και αν δεχθούμε τη συμμετοχή σε ένα συλλογικό σύστημα, ή αντιφάσει σε ένα πρότυπο, ρυθμιστικό, ανοιχτό, παραμένουν με το ίδιο άρθρο, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε την απαγόρευση άμεση ή ε, έμεσου συνδέσμου ε, με την πληρωμή. Επομένω, στην παράγραφο 3 απαγορεύουμε, επιτρέπουμε κάτι το οποίο έχουμε απαγορεύσει στην παράγραφο 2. Περιστρεφόμενες πόρτες, revolving doors, όπως είπα είναι περιορισμένη εντολή μου και άρα πρέπει να συζητήσω με τον Επιτροπό μου αν ε, μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, αλλά ίσως η περίοδος των δύο ετών να είναι υπερβολικά μακρά. θα μπορούσε να μειωθεί ίσως και σε έναν χρόνο, αλλά αυτό πάντα, όπως είπα, πρέπει να συζητηθεί πρώτα με την πολιτική μας ηγεσία. Ένα άλλο θέμα που ε, ετέθη ανταγωνισμός δηλαδή μεταξύ των ανεξαρτήτων συστημάτων. Εδώ με την ευκαιρία των ρυθμιστικών τεχνικών προδιαγραφών. Δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε. Από την άλλη όμως υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που ακριβώς προσφέρουν αυτή ε, τη δυνατότητα για την ε, εξυπηρέτηση του στόχου της καινοτομία. Όταν λοιπόν δεν είναι κατακόρυφα ενοποιημένες οι δραστηριότητες, υπάρχουν κανόνες από τον ανταγωνισμό που ασφαλώς καλύπτουν και την καινοτομία. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριος Χόμπριχ για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Απαντώντας στην πρόταση που έκανε μόλις η Κομισιόν να μειωθεί ο αριθμός των ετών από τα δύο στο 1, θα το χαιρετίζαμε αυτό, διότι θα εφαρμοζόταν με την δική μου πρόταση. Ο λόγος που εμείς επιλέξαμε αυτόν τον αριθμό ετών ε, δεν ήταν ε, και σχετίζεται με αυτό που είπατε κι εσείς ο λόγος λοιπόν που επιλέξαμε σε αυτόν τον αριθμό είναι ότι εξετάσαμε και άλλες οδηγίες για να δούμε τι είδου απαγορεύσει ισχύουν σε άλλους τομείς από άλλες οδηγίες και είδαμε για παράδειγμα στο, στον τομέα των, ε, των ελέγχων, του auditing ε, είναι κανόνας αυτός ο, ο, ένας χρόνος πέραν από κάποιες πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και γι' αυτό θεωρούμε ότι και εδώ πρέπει να ισχύσει αυτή η περίοδος του ενός έτους. Όσον αφορά τα σχόλια που κάνατε, νομίζω ότι η διαφωνία η δική σας αφορά στο τι τελικά είναι η ανεξαρτησία σε αυτό το πλαίσιο. Δεν υπάρχει ορισμός στον κανονισμό. Εξετάσαμε τα πάντα, τις ατολογικές σκέψεις. Υπάρχουν διάφορες υπόνοιες. Περιγράφεται ε, υπάρχουν διάφορες ιδέες, αλλά δεν υπάρχει ορισμός με την παραδοσιακή έννοια. Γι' αυτό και επειδή ακριβώς η εντολή μας αφορούσε και το να ορίσουμε τι είναι η ανεξαρτησία και δεδομένου ότι πρόκειται για πέτηση που άλλοτε είναι σκληρότερη, άλλοτε είναι υπιότερη. Εμείς λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν αποκλίνουμε από το κείμενο επίπεδου 1, ε, καθώς δεν δίνεται ορισμός στο επίπεδο 1. Ε, έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να, να ορίσουμε τι σημαίνει ε, όρος σαφή και αντικειμενικά κριτήρια. Η Κομισιόν πρότεινε την αφαίρεση αυτών. Εμείς όμως επιμένουμε στην επαναπροσθήκη αυτών των στοιχείων. Ε, αν δεν θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική, έχουμε και άλλες προτάσεις να κάνουμε. Και κάτι τελευταίο, η Κομισιόν αναφέρθηκε στις κατευθύνσεις γραμμές της. Όσον αφορά το δίκαιο περί αντιαγωνισμού. Δεν ξέρω αν αυτά είναι, αν ε, αυτά τα, αυτές οι νομικές πράξεις ε, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο νομικά με, το, με, το ένα, με ένα πρότυπο. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτού του είδους, αυτού του είδους τα πρότυπα θα ήταν νομικά δεσμευτικά για τους ε, παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να δω που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Δεν μπορώ να ψήσω ψήσω παραπάνω. Αυτό που θα πω είναι ότι περιμένουμε με ανυπομονησία για την επίσημη δημοσίευση, η οποία πιστεύω θα γίνει τον Ιούλιο. δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη πληροφορία σχετικά. Το χρονοδιάγραμμα είναι Σεπτέμβριος για την ε, υιοθέτηση. Ωραία. Καλές διακοπές λοιπόν και εσείς καλές διακοπές και μετά θα τα πούμε το Σεπτέμβριο. Ωραία, σας εύχομαι και εγώ καλές διακοπές, παρόλο που ξέρω πως θα πρέπει να κλείσετε και το θέμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσει λοιπόν και η διαδικασία εξέτασης, αλλά θα πρέπει να θυμόσαστε πως εμείς έχουμε την πλειοψηφία να απορρίψουμε, γιατί εκπροσωπούμε εδώ τις δύο μεγαλύτερες ομάδες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Μπορώ να περάσω στο 17, διάφορα, τίποτα. Δεν βλέπω να σηκώνονται τα χέρια που θέλουν να προσθέσουν θέματα στα διάφορα. Τρίτη 11 Ιουλίου, 9 με 12.30 και 3 με 6.30 είναι η επόμενη μας συνάντηση. Και η συνεδρίαση λύεται.